Γεια σας, συνεχίζουμε αμέσως τη συζήτησή μας. Τα χαιρετιστήκαμε, τα είπαμε. Πάμε αμέσως στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησής μας. Δηλαδή, πώ μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμών και των υπηρεσιών που ασχολούνται με την καταβλήση του οργανωμένου εγκλήματο στην Ιταλία και όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ιταλικών αρχών με του διάφορου συνομιλητέ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνέ επίπεδο όμω Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη σύνοδο από τον Εθνικό Εισαγγελέα Επεύθυνο για τα καταπολέμηση τη μαφίας, τον Πιέρο Γκράσιο, η εισαγγελία εθνική είναι ο φορέα, ο δικαστικό, ο Ιταλικό που συντονίζει τι έρευνε που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα για την καταπολέμηση τη μαφία στην Ιταλία και ζητώ από τον κύριο Εισαγγελέα να κάνει μια παρουσίαση όσον αφορά το θέμα τη συνεργασία μεταξύ των θεσμών και των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, την καταπολέμηση τη μαφία και αν μπορεί να μας πει πως οι Ιταλικές αρχές συνεργάζονται με, τις, με τους ομόλογους ε, ε, εταίρους τους σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό για να αντισταχθούν στο φαινόμενο της μαφίας. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή μετά την παρέμβαση, την παρουσίαση από την εισαγγελία του κ. Γκράσο, θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές, αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο στον εισαγγελέα τον κύριο Γκράσο και μετά θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων αν θα έχουμε χρόνο σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας κύριε Ισαγγελέφ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την παρέμβασή μου πριν να απευθύνω μια συγκεκριμένη σκέψη προς τον Τζοβάνι Φαλκόνε που ήταν ο δικαστής που δολοφονήθηκε από τη μαφία το 92 που είχε εντοπίσει στη διεθνή συνεργασία το μόνο τρόπο για να ξεκινήσει μια αποτελεσματική και συγκεκριμένη δράση γενική κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε υπερεθνικό επίπεδο και με μεγάλη συγκίνηση με σήμερα μπροστά σας σε αυτή την Επιτροπή που αποτελεί μετά από τόσα χρόνια, τόσα χρόνια μαχών και τόσων φόνων ε, το επιστέγασμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ονείρου που δεν μπόρεσε να υλοποιήσει ο Φαλκόνε, δηλαδή την απαρχή μιας ε, διαδρομής που οδηγεί σε μια πιο γενική παγκόσμια αξιολόγηση του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό ε, μεγαλύτερη εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών. Σήμερα, σαν Εθνικός Εισαγγελέας υπεύθυνο για την καταπολέμηση της μαφίας, παρακολουθώντας την εξέλιξη των εγκληματικών φαινομένων, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και να πω ότι ο Φαλκόνε ήταν ε, ήταν ένας ε, περίφημος εξαιρετικός ε, προφήτης που δεν εισακούστηκε. Είδαμε ότι οι παραδοσιακές οργανώσεις του τύπου μαφίας που υπάρχουν στην Ιταλία, όπως είναι η Κόζα Νόστρα στη Σικελία, η Καμόρα στην Νάπολη και στην Καμπανία, η στο Ιγκαλαβρία, παρόλο που παραμένουν συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη περιοχή τους, περιοχή στην οποία έχουν μεγάλο έλεγχο, σταδιακά διεύρυναν τις ζώνες επιρροής τους, εκμεταλλευόμενες μια σειρά νέων ευκαιριών που προσφέρονται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση και από την διάδοση της τεχνολογίας, ε, συσφίγγοντας διάφορες συμμαχίες με εγκριματικές ομάδες άλλων χωρών, όπως παραδείγματος χάρη με, τη, με τα κολομβιανά και μεξικανικά καρτέλ, την Κοζανόστρα, την Αμερικανική, την τουρκική μαφία, τη ρωσική μαφία, την Ιγυριανή μαφία, την αλβανική μαφία και άλλα σχήματα και μορφώματα εγκληματικά της Ανατολικής Ευρώπης, από τη Σερβία, από το Κόσοβο και από αλλού. Ε, όλες, όλη αυτή η εγκληματικότητα, όλες τις ομάδες φαίνεται ότι εντάσσονται όλο και περισσότερο, έτσι δείχνουν οι έρευνές μας σε ένα οργανικό σύστημα εγκληματικών δικτύων που συνδέονται μέσω σταθερών συμφωνιών για να χειρίζονται τις κοινέ τους παράνομες υποθέσεις για να συντονίσουν έτσι την χρήση του χρήματος των ανθρώπων και των μέσων ε, κάνοντας και συμφωνίες μη επίθεσης μη βίας, εκμεταβόμενοι αγορές και ζώνες επιρροή, αλλά όχι μόνο στα επίπεδα της παραδοσιακής ε, διακίνησης ναρκωτικών ή ε, ξεπλήματος χρήματος, αλλά χρησιμοποιώντα και κάθε άλλη εγκληματική ε, δυνατότητα που προσφέρεται σήμερα σε διεθνές επίπεδο. Οι μαφίες αυτές καθοδηγούνται από κάθε αλλαγή και τάση γεωπολιτικών παραγόντων προσπαθώντας να βρουν πιο εύκολο κέρδος και ταυτόχρονα καταλήγουν να επηρεάζουν ε, άμεσα ή έμεσα τις ίδιες τις ε, διαδικασίες τις γεωπολιτικές. Το οργανωμένο έγκλημα, το σύγχρονο, ε, παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών σε ενδεχόμενους πελάτες και από αυτή την έποψη δεν διαφοροποιείται πολύ από μια κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνδέονται ε, με παράνομη χορηγία αγαθών και υπηρεσιών, παροχή αγαθών και υπηρεσιών και στρέφονται προς τη ζήτηση ε, και η ζήτηση είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες ε, γύρω από τον οποίο στρέφονται αυτές οι δομές οι παράνομες. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος μοιάζει όλο και περισσότερο με εμπορική επιχείρηση υπερεθνική, διεθνή, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλό εμπόριο, δηλαδή την ταυτόχρονη ε, παροχή διαφόρων ειδών αγαθών και υπηρεσιών παρανόμων. Ε, πολύ συχνά δουλεμπόριο που ξεκινά από εμπόριο ναρκωτικών και μετά πάμε σε εκρηκτικά και όπλα. Στις πιο πρόσφατες έρευνες ε, φαίνεται να διαφαίνεται ένα καινούριο στοιχείο, αναδύεται, οι μεγάλες ε, οργανώσεις που έχουν παραδοσιακή ιεραρχική δομή, όπως οι Ιταλικές ομάδες, ανέπτυξαν λόγω των πιέσεων από πλευράς δυνάμεων της τάξης μια ε, ευελιξία επιχειρησιακή που χαρακτηρίζεται από μικρά δίκτυα Δηλαδή κάποιε κυψελίδε αν θέλετε τέτοια δομή, κάτι παρόμοιο με μονάδε όπω οι τρομοκρατικές ομάδε που απαρτίζονται από ελάχιστο ε, τρία άτομα και το πολύ πέντε άτομα με ε, στεγανά και μυστικότητα στον αφαντιστήριο. Είναι απομονωμένοι αυτοί οι θύλακε. Αυτό το σύστημα των δικτύων ατόμων που μετά από μία επιχείρηση ε, διαλύονται και αντικαθίσταντο συχνά χωρίς να αφήσουν ίχνη είναι κάτι που εγγυάται την συνέχεια του εμπορίου χωρίς ε, κανένα κίνδυνο για την αγορά και για την ε, εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από αυτό, ακόμα και σε περίπτωση σύλληψης ε, κάποιων από αυτά τα μέλη. Και γι' αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε να χτυπάμε ανεξάρτητα τις ομάδες αυτές τις εγκληματικές που είναι στην κορυφή αυτής της διοργάνωσης. Το κέρδος είναι τόσο ισχυρό κίνητρο σήμερα όσο σαν να είναι μια θρησκεία. Τα δίκτυα των ναρκωτικών χωρίς πατρίδα και χωρίς σύνορα αλλάζουν ε, στον κόσμο περισσότερο από ότι οι τρομοκράτες. Αλλά ο κόσμος ε, φαίνεται ότι δεν το έχει ε, συνειδητοποιήσει. Κάθε παράνομη δραστηριότητα παράγει χρήμα που ανακυκλώνεται μέρη, ξεπλένεται το κέρδος, το χρήμα είναι ο λόγος ύπαρξης του οργανωμένου εγκλήματος και ε, το να τους το πάρει το, το, το χρήμα είναι η λύση, αλλά να το βρει το χρήμα είναι το πρόβλημα. Η οικονομική κρίση και κυρίως η ρευστότητα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις που συνεχίζουν να διαθέτουν τεράστιες ροές ε, φρέσκου χρήματος και να το σπέρνουν πέρα από το παραδοσιακό εμπόριο πέρα από αυτά που αναφέραμε ναρκωτικά και όπλα, ε, σε νέες αγορές ε, που επιτρέπουν ε, σημαντικά κέρδη με μικρότερους κινδύνους για μεγάλες κυρώσεις διότι δεν τιμωρούνται επαρκώς διάφορες χώρες. Πιθανόν διότι πρόκειται περί νέου εμπορίου όπως είναι το δουλεμπόριο ε, εμπόριο ε, ε, εμπορευμάτων, παραποιημένων φαρμάκων, επικινδύνων αποβλήτων, έργων τέχνης, φυσικών πόρων και πιο πρόσφατα έχουμε φαινόμενα κλιματικά όπως είναι στον κυβερνοχώρο και η πειρατεία στις θάλασσες. Ενώ η σοβαρή κρίση του νομικού συστήματος και του νόμιμου, μάλλον της νόμιμης πίστοσης του χρηματοστικού τομέα ε, οδηγεί στην, στο να θησαυρίζουν οδηγεί στη μεγάλη τοκογλυφία και εκμετάλλευση μικρομεσών επιχειρήσεων, επίσης που πολύ συχνά ε, είναι η βασική δομή των παραγωγικών συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια η καταπολέμηση των διεθνών αυτών κλιματικών οργανώσεων στην Ιταλία ε, υλοποιήθηκε ε, με την επίθεση που κάναμε κατά των παρανόμων περιουσιών μέσω κατάσχεσης, κράτησης και ε, εντός της ποινική διαδικασίας και εκτός της ποινική διαδικασίας μέσα σε ένα καθεστώς προληπτικό πρόληψης που εφαρμόζουμε για να αντιμετωπίσουν περισσότερο τον κίνδυνο για την κοινωνία ε, και έχουμε και τα δύο συστήματα που εφαρμόζουμε και της πρόληψης ε, κινδύνου για την κοινωνία και της κατάσχεσης της περιουσίας μετά από την ποινική καταδίκη που επιβάλλεται. Τα επιτευθέντα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και λόγω ενός ε, νόμου που έδωσε τη δυνατότητα στην υπηρεσία μου, στη Γενική Διεύθυνση κατά της Μαφίας, να προβεί σε συντονισμό και των ερευνών που αφορούν τις περιουσίες τους. Κατασχέθηκαν από αδυνάμεις της αστυνομίας τα τελευταία 3,5 χρόνια ε, κινητή και ακίνητη περιουσία εταιρείε επιχειρήσεις αξίας που ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και κατασχέθηκαν αγαθά αξίας πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα στην Ιταλία μέσω μιας εθνικής υπηρεσίας που δημιουργήθηκε πρόσφατα, αυτά τα χρήματα θα πάνε σε κοινωνικά έργα. Είναι μεγάλη ηθική αλλαγή, δηλαδή επιστρέφεται στον πληθυσμό το χρήμα μέσω κοινωνικών υπηρεσιών, ε, μέσω χρήσεως από τις πλευράς των διαφόρων ε, θεσμών και των διαφόρων συνεταιρισμών των οργανώσεων για τους νέους, τα χρήματα αυτά που είχαν αφαιρεθεί από τη μαφία, από την κοινότητα, από την κοινωνία τα από ποσά σε μετρητό ή σε τρέχοντες λογαριασμούς, σε τίτλους και μετοχές αξίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, κατατέθηκαν σε ένα ενίο ταμείο για τη δικαιοσύνη και ένα κομμάτι αυτών των πόρων ε, διαιρείται σε εξίσου μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ακριβώς για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος δημιουργώντας ένα ε, θετικό κύκλο ε, μέσω του οποίου σε περίπτωση κρίσης προσπαθούμε να βρούμε ε, πόρους για να συνεχίσουμε άνευ ουδεμίας επιβραδύνσεως στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Έναντι νέων διόδων μεταφοράς των χρημάτων που ανακαλύπτονται συνέχεια είναι όλο και πιο προχωρημένες οι τεχνικές απόκρυψεις που χρησιμοποιούνται το, το παγκόσμιο χρηματοστικό σύστημα που βρήθη ε, φορολογικών παραδείσων και τραπεζικών παραδείσων δείχνει πόσο εύθραυστο είναι ε, και ε, γίνεται ένα θύλακα της ανακύκλωσης, του ξεπλήματος χρήματος. Το οργανωμένο έγκλημα άλλαξε διαστάσεις, αποκτώντας μακροοικονομικές διαστάσεις, κατακτώντας μια εμβέλεια παράνομη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παράνομα προϊόντα παράγονται σε μια ήπειρο, μεταφέρονται και διακινούνται σε μια άλλη ήπειρο και μετά καταναλώνονται ή πολλούνται σε μια τρίτη ήπειρο. Οι αποδείξεις και οι ενδείξεις τέτοιων περίπλοκων εγκληματικών φαινομένων ε, είναι διάσπαρτα σε διάφορες χώρες παραγωγής, διέλευσης, κατανάλωσης των διαφόρων ουσιών που διακινούνται. Γι' αυτό είναι προφανές ότι χωρίς μια συνεργασία, πλήρη συνεργασία που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και χρησιμοποιεί τα νομικά μέσα που ήδη έχουν δοκιμαστεί για συντονισμένη εφαρμογή και διενέργεια ε, κοινών ερευνών δεν θα καταλήξει σε κανένα σοβαρό αποτέλεσμα. Στην Ιταλία η προσπάθεια για αποτελεσματική αντίσταση κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι συνεχής έχουμε μια νομοθεσία εσωτερική από τις πιο πλήρεις και αποτελεσματικές, αλλά δυστυχώς ε, δεν καταφέρνουμε πάντα να πετύχουμε επαρκή ε, συνεργασία από πλευράς άλλων χωρών. Ε, πιστεύω πάντα ότι έχουμε συμβάλει στο να παράγουμε ένα δηλητήριο που είναι το οργανωμένο έγκλημα. Βρήκαμε το αντίδοτο, αλλά δεν καταφέρνουμε να το κάνουμε να το χρησιμοποιήσουν οι άλλες χώρες. Τώρα πια ε, δεν είναι περισσότερες χώρες με εγκληματικότητα, αλλά εγκληματικότητα, ε, υπάρχει εγκληματικότητα κολλής χώρες. Η διαφορά μεταξύ των ποινικών διαδικασιών ε, ανοίγουν ανέλπιστα κενά που τα εκμεταλλεύονται οι εγκληματικέ οργανώσει για τους μαφιόζου και εκείνου που διακινούν τα ναρκωτικά και καταστρέφουν τι νέε μα γενιές δεν μπορεί να υπάρχει στον κόσμο ένας εύκολος δρόμος διαφυγής ή χώρες που να εγγυούνται την ατιμορρησία για αυτούς. Πιστεύουμε ότι όπως και οι εγκληματίες δεν έχουν πια σύνορα για το παράνομο εμπόριό τους, έτσι θα πρέπει να κινηθούν και οι χώρες για συγκεκριμένη και αποτελεσματική ε, δικαστική συνεργασία. Ε, παραμένει ακόμα πράγματι ατελής η παγκοσμιοποίηση ε, των συστημάτων των νομικών των νομικών συστημάτων. Η προθυμένη φύση της Ιταλικής νομοθεσίας όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα ε, συνδέει όπως, όπως αναφέρθηκε ε, με την πρόβλεψη κάποιων πράξεων που διαπράττονται που, που, που δείχνουν κάποια στοιχεία ότι διαπράττονται και πιο γενικά φαινόμενα όπως είναι τα, τα, τα ομαδικά εγκλήματα, όπως το 416α το άρθρο που αναφέρεται στην ε, ομάδα ε, μαφιόζικου τύπου ή την δημιουργία ομάδας για να διαπράξει αδικήματα. Αυτή η εμπειρία μας προφανώς θα πρέπει να προσαρμοστεί με την πραγματικότητα της Ευρώπης, όσον αφορά την εγκληματικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμόσουμε και να υιοθετήσουμε κατά την άποψή μου ένα μοντέλο τέτοιου εγκλήματος ομαδικού που μπορούμε να υποθέσουμε σε ποια οργανωμένη ομάδα μπορεί να ανήκει σύμφωνα με τη σύμβαση του Παλέρμο του 2000. Πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα και η ιδιαιτερότητα και ε, το ότι ισχύει στη διεθνή εικόνα το ιταλικό σχήμα, δηλαδή του συντονισμού σε κεντρικό επίπεδο των ερευνών για το οργανωμένο έγκλημα, έρευνα από τη διενεργεί ένας φορέας όπως είναι η οργάνωση καταπολέμησης μαφίας την οποία διευθύνω, που έχει μια θέση υποστήριξης και εξορθολογισμού και αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων, διότι στην Ιταλία διευθύνει η δικαστική αρχή τις, ε, τις, αρχές, τις ε, αστυνομικές αρχές που ενεργούν τις έρευνες. Είναι ένα σύστημα που είναι μερικός κεντρικό και διατηρεί την ευθύνη των ερευνών που είναι καλό και για το έλεγχο της χώρας στις διάφορες ε, τοπικές ε, αρχές αλλά προβλέπει και κάποια όμως κεντρική, κάποιο κεντρικό συντονισμό σε κάποια φάση και με δεσμευτικά προνόμια σε περίπτωση ελλείψεων στις έρευνας ή ε, στην περίπτωση έλλειψης συντονισμού στις έρευνες που διενεργούνται. Δυστυχώς χρειάζεται να ε, λάβουμε υπόψη μας ότι απομένει προφανής δυσανάλογη προσέγγιση. Δηλαδή, πλούτος και περίπλοκος χαρακτήρας του νόμου και του διεθνούς δικαίου από τη μια πλευρά, διεθνείς συμβάσεις, αποφάσεις πλαίσια κλπ ε, μέσα υπείου νόμου soft law όπως οι συστάσεις της ΓΚΑΦΗ ε, που αποτέλεσε αντικείμενο νέας αναθεώρησης πρόσφατα το μήνα Φεβρουάριο του 2012 και που με αφηρημένο τρόπο χρησιμοποιούνται κατά της διαφθοράς του ξεπλήματος χρήματος και του διασυνοριακού εγκλήματος. Και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε νευραλγικούς τομείς δηλαδή όπως είναι η πρόληψη και η καταστολή και σώρευση των παρανόμων ε, πόρων είναι που είχαν αποτελέσματα. Τι εκτιμήσεις των διεθνών οργανώσεων τα αποτελέσματα ε, δεν είναι καθόλου ανάλογα σε σχέση με την νομοθεσία η οποία ε, έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάρια είναι, τα, είναι διάφορα τα θέματα, συγγνώμη, όσον αφορά αυτή τη διαφορά. Θα αναφερθώ σε αυτά συνοπτικά και θα σας αφήσω το πλήρες έγγραφο εδώ στην Επιτροπή, ούτω ώστε ε, να μπορείτε να δείτε καλύτερα τους λόγους ε, για αυτά, αυτά τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του συστήματος. Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα και μια δυσκολία όσον αφορά την ε, μορφή την έγκαιρη συνεργασία σε εθνές επίπεδο για τον εντοπισμό της περιουσίας αυτών οργανώσεων στο εξωτερικό για την ανάπτυξη γρήγορων ερευνών τραπεζικών. Ε, παραδείγματος χάρη, είδαμε ότι λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ένα σύστημα ε, κεντρικό για να ελέγχουν ε, ε, του τραπεζικού λογαριασμού και τι περιουσίε σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται μια δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα και ίσω να είναι σημαντικό να επιτεθεί κάτι τέτοιο. Και υπάρχει ανεπαρκή ε, ενσωμάτωση στα εφίσταμενα μέσα για την κατάσχεση των διατάξεων των κρατών μελών. Δεν υπάρχει στην ένωμη τάξη των κρατών μελών. 19 ε, από τα 27 κράτη-μέλη έχουν κάνει ενσωματώσει τι ευρωπαϊκέ διατάξει στη δική του ενόμη τάξη. Και αυτή η ατελή ε, εφαρμογή ε, δημιουργεί αβεβαιότητα όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο και είναι κάτι που δυσκολεύει την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Μετά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα των εθνικών νομοθεσιών και σε περιπτώσει κατά τις οποίες ε, έχουν ε, γίνει σωστά οι μεταφορές των ευρωπαϊκών διατάξεων στην Εθνική Ενόμη Τάξη. Διότι άμα λείπει η αρχή της αμοιβαία ε, αναγνώρισης χωρίς όρια και μετά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις από τη μία χώρα στην άλλη. Λοιπόν, όλα αυτά συνεπιφέρουν προβλήματα οδηγούν σαν αποτελεσματικότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται και, και οδηγούν και σε συνέπειες παράξενες. Σχεδόν όλες οι χώρες που θα χάρη την κατάσχεση ε, ή αντιστοιχεία αυτή της κατάσχεσης. Δηλαδή ε, μπορούν να κινηθούν και κατά τα περιουσιών όπου καταδικασμένος Κατάσταση αυτό ακόμα και αν δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση στη χώρα που έχει διαπραχτεί το έγκλημα. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η έλλειψη δίωξη και να γίνει έρευνα για εξέρευση των αγαθών ε, σε άλλες χώρες, εκεί είναι το πρόβλημα. Να γίνεται νόμιμη έρευνα και αυτό σε άλλε χώρες για να βρεθούν ε, περιουσιακά στοιχεία του εγκληματία. θα έπρεπε να μπορεί κανείς να ερευνήσει και στα άλλη χώρα ε, και αυτό είναι επιζήμιο για όλους τους πολίτες που δεν μπορεί να γίνει πλήρης έρευνα άμα κινηθεί ο εγκληματίας από μια χώρα σε άλλη. Λοιπόν, χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Ε, δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο σαν μια υποχρέωση για τις χώρες, αλλά είναι μια μεγάλη δυνατότητα και είναι κάτι πάρα πολύ καλό για να μπορέσουν να εκριζωθούν οι εγκληματικές ε, οργανώσεις από διάφορα κράτη σε μια προοπτική που βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης, της διεθνούς αλληλεγγύης και του, της κοινή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Απαιτείται λοιπόν ανανεωμένη προσπάθεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ούτω ώστε η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο να γίνει μια προτεραιότητα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήταν ευθεία παρέμβαση που θα είχε αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα οι πολλές προτάσεις ε, θα πρέπει να έχουν τελικά κοινό στόχο να ε, καταπολεμήσουμε το ρίζωμα του οργανωμένου εγκλήματος, σταθεροποίηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ήδη προτάσεις που ακολουθούν αυτή τη γραμμή, όπως ε, η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάσχεση των προϊόντων εγκλημάτων που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η προπτική μιας οδηγίας όσον αφορά το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να... η Επιτροπή μάλλον αυτή να μπορεί να συμβάλλει ούτω ώστε να καταλήξουμε σε κάποια θέσπιση κάποιων νομοθετικών μέτρων που θα μπορούσαν να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και άλλη βασική διεκδίκηση είναι η έγκριση μέτρων για αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης διαφθοράς και κυρίως της διαφθοράς με, ε, μεταξύ ατόμων ε, θα πρέπει να είναι ε, κάτι που θα είναι σε κοινή, μια κοινή αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει δράση για να εφαρμοστούν όλες οι δεσμεύσεις εφαρμογής των υφισταμένων μέτρων αυτό μπορεί να γίνει σε όλες τις χώρες, αλλά η Ιταλία είναι η πρώτη η οποία θα πρέπει να επιδιώξει να εγκρίνει το ταχύτερο ε, στην ομοθεσία της διάφορες ευρωπαϊκές διατάξεις που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην Εθνική Ενόμη Τάξη της Ιταλίας. Συνεπώς, η αποτελεσματική η αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος περνά μέσω των νέων προπτικών αυτών, αλλά θα πρέπει να μην επιδεινώσουμε και τα εφιστάμενα μέσα που υπάρχουν, όπως το καθεστώς για το data retention, για την κάτση των στοιχείων και την οδηγία Φρατίνη για τη διατήρηση των ε, ε, προϊόντων των υποκλοπών της παραγωγής των τηλεφωνημάτων. Ακούγεται ότι μπορεί να μειωθεί ο χρόνος διατήρησης αυτών των στοιχείων ε, στην Ιταλία ακούγεται ότι θέλουν να μειωθεί ε, σε έξι μήνες. Ε, αυτό δυσκολεύει τη δουλειά μου της αστυνομίας δικαστικής. Αυτή η προπτική θα είναι καταστροφή για την αποτελεσματικότητα της έρευνας όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, διότι περιορίζεται σημαντικά η ερευνητική δραστηριότητα με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα ήρθε η στιγμή, βλέποντας την σοβαρότητα του κινδύνου, οι δηλώσει των προθέσεων να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες πράξεις, ούτω ώστε η διεθνής κοινότητα, σαν ένας άνθρωπος, σεβόμενη τα δικαιώματα, το δίκαιο και τις ε, παγκόσμια αναγνωρισμένες αρχές, να μπορεί να αντισταθεί στις επιθέσεις των εγκληματίων που δεν έχουν κανένα δισταγμό, δεν έχουν καμία πίστη, δεν έχουν καμία πατρίδα, που θέτουν εν κινδύνο το μέλλον του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελέφ για αυτή την παρουσίασή σας. Θα δώσω αμέσως το λόγο στους συντονιστές για δύο λεπτά ο καθένας, ξεκινώντας από τον κύριο Ματία για, από το ΕΛΚ. Κυρία Ματία, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελέφ που απαντήσατε στην πρόσκλησή μας. Ανταποκριθήκατε και ε, για τη μακροσκελέστατη σας παρουσίαση και τη δράση σας επί τόπου. Έχω δύο ερωτήσεις κύριε Σαγγελέφ. Η πρώτη αφορά τα σίδαρα. Σε σχέση και με τους πρωινούς ε, ομιλητές που μας μίλησαν για διακίνηση ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική ή ο κύριος Μπρέιρ Ράιτ που μας μίλησε για λαθρεμπόριο όπλων από τα Βαλκάνια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο την άποψή σας για το θέμα των συνόρων. Κατά τη γνώμη σας, τα σύνορα που δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί στο ιστορικό της Ένωσης δεν έχουμε σύνορα. Αυτό τι επίπτωση έχει στην εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στο εσωτερικό της Ένωσης ή δεν έχει. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι το οργανωμένο έγκλημα ε, δρά και έχει τον ίδιο αντίκτυπο και εκτός της Ένωσης και εντός της Ένωσης, δηλαδή και έξω θέν και στο εσωτερικό. Είναι θέμα συνόρων και τα καλύτερα αποτελέσματα στις έρευνες των διοκτικών αρχών που φτάνουν σε εσά πολύ συγκεκριμένα. Ε, γίνονται σε διμερή συνεργασία από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ή ε, είναι καλύτερα τα αποτελέσματα κατόπιν συνεργασίας ε, των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων Eurojust ή Europol. Θα ήθελα την άποψή σας παρακαλώ ως κάποιου που ασχολείται καθημερινά με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κροτσέτα. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελέφ που είσαστε εδώ μαζί μας. Οι παρεμβάσεις σας σας έχουμε δει αλλες δυο δύο-τρεις φορές και μας βοήθησαν οι παρεμβάσεις σας στο παρελθόν να δημιουργήσουμε τις, να σχηματίσουμε τις εργασίες τη Επιτροπή αυτή, στην οποία συζητούμε. Σε κάποιο σημείο μιλήσατε για γεωπολιτικές διαδικασίες που ενδιαφέρουν τις εγκληματικέ οργανώσεις. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται περαιτέρω ευάθυνση από αυτών των πτυχών, διότι πολύ συχνά όταν γίνεται λόγος για τη διάδοση των εγκληματικών οργανών στον κόσμο, ε, πολύ συχνά θεωρεί κανείς ότι η, εγκληματική, η μαφία από την Καλαβρία της Σικελία θα κατακτήσουν όλη την Ήπειρο. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, πράγματος χάρη, να θεωρήσει κανείς το ότι είναι τόσο ισχυρέ αυτέ οι μαφίε που έχουν δημιουργήσει ένα μοντέλο αναφοράς ε, και, και παρόλο που είναι σύγχρονος ότι μπορούν να οργανωθούν σε τέτοιο επίπεδο τόσο μεγάλο εμπόριο και κυκλοφορία. Θα ήθελα να ξέρω, κατά την άποψή σας από ερευνητική σκοπιά, Ξέρουμε για οργανώσεις που είναι οργανωμένες σε διάφορες χώρες. Ανατολική Ευρώπη. Όμως πέρα από την Ανατολική Ευρώπη, που είναι από τα θέματα που συζητάμε συχνά, πώς λειτουργούν αυτές οι εργαματικές οργανώσεις στις ζώνες που αποκαλούνται ε, αθώς, ότι δεν υποψιάζεται κανείς ότι δράει η, ε, η μαφία, όπως η Δυτική Ευρώπη, Γερμανία, πώς λειτουργούν, στο Βέλγιο, πώς λειτουργούν. Καταλαβαίνω ότι σας κάνω μια ερώτηση που μπορεί να οδηγήσει σε ολόκληρη εργασία για την ε, σύγχρονη κλιματικότητα. Αλλά είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε πώς είναι οργανωμένες αυτές οι οργανώσεις στην Ευρώπη. Για να δούμε πιο ακριβώς, πιο επακριβώς τι είδους δουλειά θέλουμε να κάνουμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Άντε ο κύριος Νιούτον Τόν. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας κύριε Σαγγελέφ και ευχαριστώ που ήρθατε. Τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει στη δουλειά σας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλατε να δείτε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα ας πούμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. FBI μήπως στην Ευρώπη για να αγωνίζεται ε, εναντίον των κακών ανά την Ευρώπη. Θέλετε κοινοτικά πρόστιμα, τα ίδια σε όλες τις χώρες, για να μην εξειδικεύονται οι κακοποιοί σε μία χώρα, γιατί είναι πολύ εύκολο να καταφύγουν εκεί. Θα θέλατε ε, ευρωπαϊκές φυλακές. Τι μας συστήνεται να συστήνουμε εμείς του χρόνου στην έκθεσή μας όταν θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Επίσης, ο κύριο Κύρκοπ από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές για δύο λεπτά πάντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από λίγα λεπτά ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ευρώπη. Πρέπει να πω ότι στα πλαίσια των συζητήσεων που κάνουμε εμείς εδώ υπάρχουν πολλά ε, σύνορα τεχνολογικά, τηλεπικοινωνιών, ποινικού δικαίου, χρηματοπιστωτικά, τραπεζικά, επαγγελματικά, ε, εργασιακά και φυσικά όλοι οι κανόνες ε, και οι νόμοι που ισχύουν ε, ε, σε εταιρείες που είναι καθόλου αξιοσέβαστες εκ πρώτης όψεως και στην επιφάνεια, αλλά από κάτω έχουμε ξέπλυμα χρήματος, πλαστογραφία, παραχάραξη και τα λοιπά, από όλους αυτούς που δρούν εγκληματικά. Συνεχίζω λοιπόν μετά από τις ερωτήσεις του κυρίου Νιούτον Ντάν και θα με ενδιαφέρει πραγματικά να μάθουμε πώς μπορούμε εσάς να σας βοηθήσουμε στη δικιά σας δουλειά σε μια συγκεκριμένη χώρα ε, με συγκεκριμένο είδος εγκληματικής δραστηριότητας και η δουλειά σας είναι πολύ δύσκολη. Θα ήθελα ειλικρινά να μάθω ακριβώς λόγω αυτών των συνόρων που όντως υπάρχουν, αλλά πολύ συχνά είναι καταφύγιο για όλους αυτούς ε, τους εγκληματίες και τις οργανώσεις, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε και σε ό,τι αφορά τούτη εδώ την Επιτροπή, γιατί ασχολείται με ένα ευρύτατο φάσμα ε, εγκληματικών ε, συμφερόντων και ενδιαφερόντων όσο και τόπων τι μπορείτε εσείς να μας προσφέρετε από την εμπειρία σας και σε εμά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Δύο λεπτά για την ΚΟΕ, ο κύριος Σόντεργαρτ, παρακαλώ. Ε, ε, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο διάφοροι οργανισμοί, διάφοροι, διάφορα θεσμικά όργανα της ε, Ιταλίας συνεργάζονται για αυτούς τους στόχους. Ε, αν τώρα ε, οι κακοί αντιμάχονται τους καλούς, είναι πάρα πολύ δύσκολη η μάχη, είναι δυσνόητα αυτά που συμβαίνουν και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Το πρόβλημα είναι όταν οι κακοί δουλεύουν για τους καλούς ε, ε, στην αστυνομία παραδείγματος χάρη. Τι γίνεται αν οι αστυνομικές αρχές ε, συνεργάζονται με τη μαφία, τι γίνεται αν δεν είναι είδα το στεγής διάφορες διοικητικές δομές όπως το δικαστικό σώμα, παραδείγματο χάρη. Σε ποιο βαθμό συμβαίνει αυτό, μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση βάσει τη εμπειρία σα ε, και ποιε ειδικέ προκλήσει πρέπει να αντιμετωπίσουμε λόγω αυτού. Ευχαριστούμε δύο λεπτά, ο Μποργέτσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς όχι μόνο επίσημα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο εισαγγελέα που είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση μαφία και για την ανάλυση που έκανε και κυρίω για τι δραστηριότητέ του. Συνεχή δραστηριότητα που ασκεί και προσφέρει έτσι στη χώρα, στη χώρα μα, αλλά και στην Ευρώπη που κοιτά με όμα ερευνητικό προς τη μεριά μας και ανήσυχο αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά την καταπολέμηση των διάφορων μορφών οργανωμένου εγκλήματος τύπου μαφίας και για τους κίνδυνου μόλυνση που υπάρχουν και διάδοση του φαινομένου. Από αυτή την έποψη πιστεύω ότι έχοντας έστω και σύντομη θεσμική εμπειρία με υπεύθυνη κυβερνητική σε ευαίσθητο τομέα όσον αφορά την κατεύθυνση της ε, μαφίας, επομιζόμενες πολιτικές και ιστορικές ευθύνες ότι πρέπει να σας ρωτήσω μήπως θεωρείτε αναγκαίο σε αυτή την ευρωπαϊκή έδρα, σε αυτό το βήμα να πείτε ξεκάθαρες κουβέντες που πλέον ε, ε, δεν καλύπτεται παρκώς όταν μέσα ενημέρωση. Το Ιταλικό κράτος ε, διαπραγματεύτηκε με τη μαφία και σε ποιο επίπεδο, σε ποιο επίπεδο είναι οι έρευνες όσον αφορά αυτό το θέμα. Ε, μπορείτε ίσως να μας δώσετε όπως και στην Ιταλική Επιτροπή της Μαφίας να δώσετε κάποια έγγραφα εμπιστευτικά για όλα αυτά τα έγγραφα να μας δοθούν για τυχόν συναλλαγές του κράτους με τη μαφία. Διότι αισθανόμαστε εμείς σαν Ιταλοί την υποχρέωση να ε, αυξήσουμε το επίπεδο της έρευνας και της επεξεργασίας ε, και θεωρούμε ότι η νομοθεσία μας είναι άριστη όσον αφορά την κίνηση που κάνει για την κατάσχεση των, ε, της περιουσίας και την εξάλληψη των περιουσιακών στοιχείων της μαφίας. Και έχει πάρα πολλές επιτυχίες όσον αφορά την αστυνομία και εξασφαλίζεται έτσι η σύλληψη επικινδύνων μαφιόζων οι οποίοι συνελήφθησαν πάνω απ' όλα πρόσφατα χάρη σε εκείνους που ήταν, ανήκαν σε αυτούς αρχικά. Ε, έχουμε λοιπόν καθήκον έναντι των άλλων χωρών μελών να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι και να προσφέρουμε και για λόγους ιστορικούς και πολιτικούς την αλήθεια. Αυτό πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει συγητήσει ο κ. Γιακολίνο για ένα δίλεπτο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρέμβαση, την ε, διαχείριση κάθαρη... του εισαγγελέα του κ. Γκράσο, ο οποίος υπογράμμισε ε, το, το, το πώς πως ε, είδαμε ένα φαινόμενο που είναι υπερεθνικό αυτό τα κέρδη των ε, οργανώσεων αυτών. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που έθεσε ο κ. Αγγελέας, όπου λέει ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει πατρίδα σήμερα. Είναι μια οργάνωση χωρίς σύνορα, άρα χωρίς ηθαγένεια. Εκφράζοντας έτσι μια κρίση ε, που επικρατεί. Ε, αναφέρατε και σωστά και δίκαια τον κύριο Φαλκόνε που εδώ και 20 χρόνια δεν φανταζόταν ότι μετά από 20 χρόνια αυτό το θέμα, το τόσο σημαντικό, επιτέλους θα αναγνωριζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, τουλάχιστον στο τέλος των εργασιών μετά από ένα χρόνο θα πρέπει να ετοιμάσουμε μια έκθεση. Σας ρωτώ, τι σκέφτεστε όσον αφορά αυτή την ε, συνεργασία, τη διεθνή, δικαστική και αστυνομική που είναι ουσιαστική για την ε, αντιμετώπιση των μαφιών και κυρίως ε, των εσόδων των παρανόμων αυτών των οργανώσεων. Τι σκέφτεστε για μια σούπερ ε, εισαγγελία ευρωπαϊκή, τι θα έπρεπε να έχει αυτή η σούπερ εισαγγελία ευρωπαϊκή για να είναι η ίδια μια προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια. Εσείς πριν αναφερθήκατε στα χαρακτηριστικά του, του αδικήματος, του εγκλήματος του ομαδικού. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια φετηρία, ούτω ώστε αυτή η μορφή εγκληματικότητας εκτός του να καλύπτεται νομικά στην Ιταλία να μπορούσε να καθορίζεται και στις άλλες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελέφ. Ευχαριστώ. Μπορσελίνο. Κυρία Μπορσελίνο, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σαγγελέφ για την ε, ανάλυση, την τόσο ξεκάθαρη και σαφή που αφορούσε την εξέλιξη των εγκληματικών αυτών φαινομένων. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ε, πριν από όλα αυτά θα πρέπει να ασχοληθούμε με την πρόληψη, να καταλάβουμε άλλα λόγια πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτά που συνέβησαν στην Ιταλία εδώ και τόσο καιρό και να μην μολύνει πλήρως ε, και την υπόλοιπη Ευρώπη αυτό το φαινόμενο αλλά το να μιλάμε απλώς για επιμόλυνση ίσως είναι κάτι επιφανειακό. Σήμερα μιλήσαμε για ένα είδος ε, Μιλήσαμε το ένα είδος άρθρου 416α ευρωπαϊκού. Μιλήσαμε για μικτές ομάδες ε, παρέμβασης. Μιλήσαμε για έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα. Με, συζητήσαμε τα προνόμια, τα όρια του. Ε, κουβεντιάσαμε πάνω απ' όλα ε, κοινού νόμους που θα επέτρεπαν τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα τεράστια κέρδη ε, του οργανωμένου εγκλήματος και μιλώντας γι' αυτό δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη σηματεία της κατάσχεσης που στην Ιταλία ε, έχει μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή ε, ηθική, ηθικό σκοπό, διότι τα κατασχεθέντα κέρδη χρησιμοποιούνται για ηθικούς σκοπούς. Δεν μπορούμε να μην το συνδέσουμε αυτό με την ιδέα της διαφθοράς, με το φαινόμενο της διαφθοράς. Και εδώ και το ερώτημά μου. Η διαφθορά που τροφοδοτείται το ΣΥΠΗΝ από τα τεράστια κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος ε, σίγουρα και το ξέρουμε καλά στην Ιταλία ε, η διαφθορά ε, τελικά οδηγεί σε παρέμβαση στην πολιτική. Τι γίνεται, αν γίνεται κάτι στην Ιταλία για να εμποδίσει τη διείσδυση της ε, μαφίας στην πολιτική. Ρωτάω για την Ιταλία, γιατί αυτό θα μπορούσε να μας το δείξει να καταλάβουμε πώς στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να καταπολέμησουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τη διείσδυση της μαφίας στην πολιτική και συνεπώς να μπορεί να επηρεάζει και τις ε, διάφορες επιλογές που γίνονται. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κυρία Βάιλερ. ich kann's ganz schnell machen. Είμαι πάρα πολύ σύντομη είπατε στην τοποθέτησή σας ότι ήδη υπάρχει από σήμερα δυνατότητα κατάσχεσης ή δίμευσης, τουλάχιστον στον τόπο που έχει γίνει η αξιόπιστη πράξη αυτή. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες επαρκούν για να αντιμετωπιστεί αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχουν χώρες που δεν ε, τις έχουν ακόμα ε, εφαρμόσει, υιοθετήσει, γιατί η δίμευση, η κατάσχεση των προϊόντων εκκλήματος είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική για να ε, προληφθούν άλλες δραστηριότητες. Μπορείτε να μας τα πείτε αυτά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. mam... Ευχαριστώ. Θα είχα ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα, κύριε Σαγγελέφη, διότι έχετε μεγάλη πρακτική εμπειρία. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νομοθετικές αρμοδιότητες. Στην ε, χώρα σας ασχολείστε επίσης με το Ιταλικό Δίκαιο και θα ήθελα να μάθω ε, το ισχύον δίκαιο ανεξαρτήτως της ε, ποιότητας του πώς ε, συνδέεται με την δράση της καταπολέμησης οργανωμένης εγκληματικότητας σε κάθε χώρα. υπάρχουν κανόνες, διατάξεις, δεν υπάρχουν νομικά κενά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όμως δεν λειτουργεί αισίως το σύστημα και άρα η ποιότητα των νομικών διατάξεων επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της οργανωμένης εγκληματικότητας. Ποια πρέπει ιδανικά να είναι η η προστιθέμενη αξία μιας ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τα οικία δίκαια. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε τώρα ο Ισαγγελέμ Γκράσο για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. <laughs> Eh, Μάλιστα, τηλεγραφικά, έτσι. Σύνορα. Τώρα πια. Ποια μπορεί να είναι τα σύνορα. Στην Ευρώπη υπάρχουν σύνορα. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε ας πούμε, έχουμε τις ακτές. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο να ελέγχουμε όλες τις ακτές. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια φίλτρα ε, στο εσωτερικό, γιατί σήμερα ε, μπορεί κανείς με ένα φουσκωτό να έρθει πάρα πολύ γρήγορα με ένα ταχύπλο στην Ευρώπη από τη θάλασσα. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει με τρόπο πολύ αυστηρό και μεθοδικό να εφαρμόζουμε αυτά για να ελέγχουμε τα σημεία εισόδου. Ε, όπως τα αναφέραμε αυτά. Επίσης, ε, έχουν περισσότερες ε, συνεργασίες, καλύτερη αποτελεσματικότητα, οι διμερείς συνεργασίες ή τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Κοιτάξτε, εξαρτάται από την αξιόπινη πράξη. Εάν είναι υπερεθνική, εντάξει. Η, ε, πολυ, πολυεθνική δεν είναι πάντα διμερής. Ε, παράλληλα ε, γίνονται έρευνες, ιδιοκτικές αρχές δρούν σε διάφορες χώρες και αυτό έχει τεράστιες επιτυχίες καμιά φορά με συλλήψεις ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες θα πρέπει επίσης ε, να ε, προλαμβάνουμε με αίτηση δικαστική συνδρομής, αστυνομίας και δικαιοσύνης για ανταλλαγή απόψεων εκ των προτέρων. Για να έχουμε και εμεί ε, την ίδια ταχύτητα με τις εγκληματικέ οργανώσεις. Αλλιώ θα είμαστε καταδικασμένοι να μένουμε πάντα πίσω, να υπολοιπόμεθα έναντι των κακοποιών και θα πρέπει να δούμε και τα μέτρα. Ε, ε, γιατί όταν φτάσουμε εμείς με τις διοκτικές αρχές έχουν εξαφανιστεί και είναι δύσκολο ε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις οργανώσεις. Περνώ αμέσω άλλες ερωτήσεις. Γεωπολιτική φύση. Θυμάμαι και θυμίζω πάντα το θέμα της πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Αμέσως μετά είχαμε μια υποκλοπή ενός τηλεφωνήματος ένας ε, μαφιόζος ήταν στην Ιταλία και ο άλλος ήταν στο Δυτικό Βερολίνο και του είπε να πας αμέσως στο Ανατολικό. Και τι να κάνω, να αγοράσεις. Αγόρασε ό,τι βρεις. Δισκοτέκ, night club, ε, ξενοδοχεία, πιτσερίες, ό,τι πωλείται πάρτο. Τα πάντα, όλα. Και την ίδια μέρα έγιναν εγκληματικές αγορές τέτοιες. Και άνοιξαν εγκληματικές αγορές καινούργιες. Η πρόληψη λοιπόν είναι να καταλαβαίνουμε πότε το οργανωμένο έγκλημα ε, θα περάσει προς ένα πιο ασθενές πολιτικό σύστημα, γιατί υπάρχουν πιο ασθενείς θεσμοί κάπου και από εκεί ε, μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση και την πολιτική και την οικονομική και την κοινωνική. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο μάλιστα, για να αποφύγουμε να υπάρξουν μαφιόζικα κράτη. Δηλαδή, εκεί που το οργανωμένο έγκλημα καταφέρνει να ε, επηρεάσει στις αποφάσεις το κράτος με τα επακόλουθα διαφθορά κτλ. η μαφία όταν κάνει business δεν ε, είναι ορατή. Έχει συγκεκριμένη στρατηγική. Σε πολλά μέρη και στη χώρα μας και στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να μετρήσει κανείς ε, ε, το οργανωμένο έγκλημα με βάση στατιστική, ανθρωποκτονίες, ξέρω εγώ, εγκλήματα τέτοια. Γιατί αυτό είναι τελείως λάθος μέτρο. Θα πρέπει να πω, αντίθετα, ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα τα πρόσωπα που φαινομενικά δεν επιδίδονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αλλά υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, νοτίτσι εκρήμινης, ενδείξεις που μας βοηθούν για να ε, προχωρήσουμε σε μία δίωξη. Και αυτό ε, σημαίνει διεθνή συνεργασία, ιδιαίτερα όταν δρούνε ε, κάποιοι σε μια άλλη χώρα και είναι πολύ γνωστοί, συσημασμένοι στη χώρα προέλευσής τους. Αυτή η σχέση που πλέον έχουμε ε, δει και στη χώρα μας ως εμπειρία μεταξύ Βορρά και Νότου είναι μια ευρύτατη συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών που κάνουν τις έρευνες και των δικαστών ε, με τη χώρα προέλευσης ορισμένων τέτοιων καταστάσεων. Πώς να το χαρακτηρίσω κάποιων όχι εθνικών αλλά εγκληματικών δραστηριοτήτων που έχουν μετατεθεί σε άλλες χώρες. Ε, για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε αυτό το φαινόμενο να αναδυθεί καν να εμφανιστεί. Ε, υπάρχει και μία τάση να αρνείται κανείς την ύπαρξη την ίδια του φαινομένου, γιατί κανείς δεν είναι πρόθυμος να δεχτεί, να παραδεχτεί ότι έχει στην επικράτειά του τέτοιο. Και αυτό είναι το πιο υποχθόνιο και το πιο ύπουλο, ε, διότι Απ' έξω δεν μπορεί κανείς, ε, είναι αδύνατο ε, προληπτικά να δράσει. Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Ε, τι εξυπηρετεί. Είναι μια νομοθεσία. Δεν μπορεί όμως να εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη με την αμοιβαία αναγνώριση. Εγώ δεν θέλω ε, ξέρω ότι είναι όνειρο να σκεφτόμαστε να υπάρχει ενιαία νομοθεσία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα με την οποία δουλεύω και ε, καλό είναι να έχει κανείς και όνειρα και να μην θεωρεί ότι είναι ουτοπία, αλλά μια ελπίδα που προσδοκεί να επαληθευτεί και να γίνει πραγματικότητα. Κοινέ φυλακές. Τι να τις κάνουμε, τις κοινοτικέ φυλακές. Ενδεχομένω ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ διαφόρων κρατών. Ε, μάλλον όχι, ε, ε, δικαστικών υπαλλήλων. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μορφή συνεργασίας. Αλλά δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες ακόμα η συνεργασία δικαστική. Ή μπορεί να υπάρχει μια πολύ σκληρή φυλακή ή ποινή φυλάκισης για να μην μπορεί ο νονός να εξακολουθεί να δρά από μέσα από τη φυλακή, είναι πιο σκληρή η κράτηση, ένα είδος απομόνωση στη φυλακή που να αποτρέπει τέτοιες ε, επιπτώσεις. Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάτι Τώρα απαντώ στον ε, Ευρω... για το, το Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Τέθη ένα ερώτημα από περισσότερον από, από έναν βουλευτές. αυτό. Δεν ε, πιστεύω στη δυνατότητα να υπάρχει ένας υπέρ εισαγγελέας Ευρωπαίος. Όχι για έναν απλούστατο λόγο. Διότι τα κράτη-μέλη να απεμπολίσουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις νομίζω ότι είναι κάτι ανέφικτο. Βλέπω έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα όμως που μπορεί να προασπίζεται πλήρως τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Αυτός ο εισαγγελέας θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο εκείνο που έχουμε στην Ιταλία, όπως το ε, Υπουργείο, στο Υπουργείο. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος από οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία. Θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να διώκει όλες τις εγκληματικές πράξεις και όλες τις ε, υποθέσεις που δικοινοποιούνται και θα πρέπει να ε, ελέγχει και να διευθύνει και την, ε, τις αστυνομικές υπηρεσίες που διενεργούν τις έρευνες. Αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο και το ενδεδειγμένο που ενδείκνεται για μια δράση, πραγματικά δράση πράσπισης συμφερόντων της κοινότητας, διότι είναι υπερεθνικά συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε σε επίπεδο ενός συστήματος που μπορεί, κατά την άποψή μου, ε, να είναι στο επίπεδο του αδικήματος αυτού της εγκληματικής πράξης σε υπερεθνικό επίπεδο. Όπως και τα σύνορα, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά σύνορα τεχνολογικά, σύνορα συμφερόντων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όχι ένα σύνορο κοινό κατά της εγκληματικότητας. Αν θέλει η βιομηχανία να προστατεύσει πραγματος χάρη το, τα πνευματικά της δικαιώματα, τη μάρκα της πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύνορο κατά του εγκλήματος, κοινό σύνορο για να καταφέρουμε να πλήξουμε τα παραποιημένα τα προϊόντα, όπου και να βρίσκονται αυτά. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε σχέσεις με χώρες όπως είναι η Κίνα, που είναι στο επίκεντρο αυτού του εμπορίου, του λαθρεμπορίου των παραποιημένων προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να έχει μια ενότητα να προσπαθήσει και από την έποψη τη διπλωματική πρώτα απ' όλα και σε διαφορετικά επίπεδα μετά να πετύχει συνεργασία και με τις χώρες που είναι εκτός Ευρώπης. Διότι σήμερα πολλά προβλήματα δεν γεννώνται στην Ευρώπη, όπως σας είπα, γεννώνται σε άλλες υπήρους και η Ευρώπη ε, είναι θύμα των προβλημάτων, όπως πολύ συχνά γίνεται και με τις επιθέσεις οικονομικές, σηματοτιστικές, όπως βλέπουμε. Τούτων λεχθέντων, πιστεύω ότι οι διάφορες υπηρεσίες που συνεργάζονται στην Ιταλία μπορούν να έχουν υποστεί ε, διεισδύσεις από τη Μαφία. Εγώ στην υπηρεσία μου, όταν ήμουν εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Παλέρμο, είχαν διεισδύσει κάποια άτομα στις αστυνομικές δυνάμεις που συνεργαζόταν με τον εχθρό με τη μαφία. Είχαμε τη δύναμη και την ικανότητα να κάνουμε να αποκαλυφθούν αυτοί και να εξαθρώσουμε αυτό το φαινόμενο και να βγάλουμε αυτόν τον καρκίνο από τη δύναμή μας. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζονται ε, ε, προσεκτικές προσεγγίσεις για να μπορούν να εντοπίζουν ο κάθε φορέας αν ε, ε, κάνει κάποια λάθη και αν αυτό οφείλεται σε αμέλεια ή προδοσία, η παρέκκληση. Αν είναι προδοσία έναντι του εχθρού που είναι το οργανωμένο έγκλημα. Αν διαπιστώνται κάποιε παρατυπίες και περίεργες κινήσει. Όσον αφορά το κύριε Μποργέσιο, ε, τις ε, Εγώ συμφωνώ με σας να ψάξουμε να βρούμε την αλήθεια. Ήδη υπενθύμησα ότι είχα το προνόμιο να δεχτώ τις δηλώσεις αυτού του συνεργάτου, Σπατούτσο λεγόταν, ε, συνεργαζόταν, συνεργάτης αστυνομίας, που ξανά άνοιξε όλο το κεφάλαιο των ερευνών. Έρευνες που όπως ξέρετε ακόμα συνεχίζονται. Όταν ολοκληρωθούν βέβαια οι έρευνες, ως παράδειγμα εκείνου που δεν πρέπει να συμβεί σε καμία χώρα του κόσμου. Διότι κανένα κράτος δεν πρέπει να, να διαπραγματεύεται με κλιματική οργάνωση. Εάν ξέρουμε θα μπορούν να είναι χρήσιμοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δοθεί αυτή η γνώση. Όμω, όπως λέει κάποιο, αφήστε μας να δουλέψουμε, αφήστε να γίνει αυτό που γίνεται δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσει με εγκληματική οργάνωση που έχει διαπράξει τέτοιε φρικαλαιότητε, τόσα εγκλήματα. Διότι έχω πάντα υπόψη μου, στο μυαλό μου, ε, αυτό που έγινε στην αυτοκινητόδρομο στο Καπάτσι, ε, όπου ανατράπηκε, εκτινάχτηκε το αυτοκίνητο με τη βόμβα, πετάχτηκε εκατάδε χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο του Φαλκόνε ε, που χτύπησε και σκοτώθηκε αυτός και η γυναίκα του ή το κτίριο στη Βία Νταμέλιο όπου βρέθηκαν ε, έγινε έκρηξη και βρέθηκαν ακόμα και κομμάτια ανθρώπων σε, ψηλά, σε ψηλούς ορόφους. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κανείς καμία σχέση με αυτούς τους εγκληματίες, με τέτοιου είδους εγκληματικότητα. Η δικαστική συνεργασία. Όσον αφορά την υπερ, τη σούπερ εισαγγελία απάντησα. Τώρα λοιπόν αυτό το αδίκημα, το έγκλημα του να δημιουργεί κανείς ομάδα για εγκληματική πράξη, το ανέφερα αυτό. Εγώ δεν είμαι για διάφορα παράνομες πράξεις που έχουν δημιουργηθεί και πραγματοποιούνται αυτά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για μαφία της Ιταλίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την ποινική ανάλυση και να ε, δούμε τι, πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Διότι το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι μόνο εγκληματικός παράγων και τελεία και παύλα. Πρέπει να τη δούμε και σαν κοινωνικό φαινόμενο, κοινωνικό γεγονός. Γιατί πολύ συχνά δίνει δουλειά η εγκληματικότητα. Είναι ένας παράγων οικονομικός. Είναι κάτι, ένας παράγων που πειράζει και την πολιτική. Η αξιολόγηση λοιπόν θα πρέπει να είναι σφαιρική και θα πρέπει να αφορά όλες τις πτυχές του φαινομένου. Και μέσω της ανάλυσης θα πρέπει να βρούμε αυτό το, την αξιόπινη πράξη που θα πρέπει να χτίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους και να μπορεί να είναι κάτι αναγνωρίσιμο, κυρίως κερμινεύσιμο και εφαρμόσιμο από τους δικαστές. Διότι το ποινικό δίκαιο και οι δίκες ε, έχουν ένα σκοπό να καταδικαστούν και οι διαδικασίες και να καταδικαστούν και οι υπεύθυνοι των πράξεων υπάρχουν και άλλες τυπολογίες αξιόπινων ε, ε, πράξεων. Κάποιος αναφέρθηκε σε εξωτερικό διαγωνισμό. Εγώ πρώτα απ' όλα θα έλεγα να έχουμε τη σύσταση συμμορίας και μετά να μπούμε σε άλλες τυπολογίες ε, αξιόπινη που είναι πιο περίπλοκη. Εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να είναι σίγουρο. Εάν υπάρχει μία συμπεριφορά που πρέπει να τιμωρείται, αυτό δεν θα πρέπει να αποφασίσει το κοινοβούλιο, θα πρέπει να παίρνει τυπική μορφή για να αποφεύγεται η ερμηνεία. Δηλαδή, να παίρνει κανείς ψήφους από εγκληματική οργάνωση είναι ε, αξιόπινη πράση. Αλλά ε, το, το κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει εάν δεν ερμηνεύεται πολύ σωστά, αν είναι αδίκημα ή όχι αυτό. Αυτή είναι η θέση μου όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα. Τώρα, εξωτερικό διαγωνισμό είναι θέμα ποινικού δικαίου, ουσιαστικού ποινικού δικαίου, που είναι πολύ ευρύτερο. Δεν μπορεί να το εξαλείψει κανεί αυτό. Όταν θέλει κανεί να τιμωρήσει μια συμπεριφορά, πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ούτω ώστε να αναγνωρίζεται μια συγκεκριμένη πράξη σαν, κάτι, σαν μια κολάσιμη πράξη και να αναγνωρίζεται από όλου. Διαφθορά και κλείνω. Δυστυχώ, βλέπετε, ε, διαφθορά υπάρχει και σχέση μαφίας με πολιτική. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στην Ιταλία υιοθετήσαμε κάποιους νόμους, κάποιες διατάξεις όπως διάλυση των κοινοτικών συμβουλίων που είναι ερετός, ερετό οργανό που εκλέγει ο λαός που με διοικητική διαταγή διαλύεται. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορούμε να έχουμε. Αλλά βέβαια με προϋποθέσεις. Θα πρέπει αυτός ο φορέας να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά λίγων ατόμων προνομιούχων, που μετά είναι, βρίσκουμε ότι είναι οι μαφιόζοι ή αυτοί που ανήκουν σε μια εγκληματική οργάνωση. Όπως ε, ανταλλαγή ψήφων, σχέσεις πολιτικών μαφίας, είναι κάτι που και εμείς ευχόμεθα να καλείται η νομοθεσία μας, διότι τώρα τιμωρείται τιμωρείται μόνο αν δίνονται ψήφοι με αντάλλαγμα χρήματα. Αυτό προβλέπει η ε, νομοθεσία μας για τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε. Και ε, ξέρουμε ότι πολλές χώρες στην Ευρώπη ε, ε, κυνηγάνε το ξέπλυμα χρήματος. Θα μπορούσαμε και εμείς να πάρουμε πολλές χώρες, νομοθεσίες, αποφάσεις πλαίσιο που δεν υιοθετήθηκαν από τη χώρα μας και επικυρωθεί. Εγώ έχω ολόκληρο κατάλογο που με φαίνει και σε δύσκολη θέση θα έλεγα. Και εδώ φαίνεται και ποιε από αυτέ τι χώρε έχουν ενσωματώσει στη δική του ένωμη τάξη αυτέ τι αποφάσει και ποιε χώρε πρέπει να το κάνουν αυτό. Σε πολλά, όσο αφορά πολλού νόμου, είναι και η Ιταλία που δεν έχει εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο στην νομοθεσία τη. Δεν αρκεί η απόφαση πλαίσιο. Το όνειρό μου είναι να έχω ένα νόμο, νόμο που να ισχύει για όλη την Ευρώπη. Πολλές χώρες πράγματι δεν έχουν σωματώσει στην ένωμη τάξη τους ε, την κατάσχεση. Ίσως δεν αντελήφθησαν ακόμα τη σημασία που έχει αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο. Είπα ότι ο μόνο σίγουρο, βέβαιο τρόπο για να χτυπήσει τι εγκληματικέ οργανώσει είναι να τι χτυπήσει στι τσέπε, στην περιουσία του. Διότι φυλακή, όποιο πάει στη φυλακή αντικαθίσταται από άλλου. Και δεν χτυπάμε έτσι όσο, όπως χτυπάμε όταν επιτεθούμε στην περιουσία τους. Αυτό είναι σημαντικότατο και έχει προτεραιότητα στην προσπάθεια καταστολής που καταβάλουμε. Κλείνω με την προστιθέμενη αξία ε, του νόμου ε, πέρα από τις διατάξεις που τιμωρούν συμπεριφορές, παραλήψεις χρειάζεται μια πρόληψη πρόληψη που είναι σημαντικότατη διότι η πρόληψη αποφεύγει το να μπούμε στην παθολογία του, της αξιόπινης πράξης. Θέλουμε ένα νόμο που να τιμωρεί πράγματι τα φαινόμενα, αυτή είναι η ιδιότητα και μετά έχουμε την πρόληψη ε, που έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στην εφαρμογή του νόμου. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί απάντησα πολύ γρήγορα ε, σε θέματα που θα χρειαζόταν εβδομάδες εμβάθυνση διαφορετικά. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελεφ, λέει Πρόεδρος. Πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο εμβαθύνατε σε αυτές τις τυχές, σε αυτά τα ζητήματα που κι εσείς όπως και οι πρωινοί ομιλητές υπογραμμίσατε κι εσείς την ανάγκη που υπάρχει για ένα νόμο, ευρωπαϊκό νόμο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα ευρωπαϊκά. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ. Μου δίνετε και τον κατάλογο των αποφάσεων που υθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και που λάβαμε τον κατάλογο. Και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες δεν έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά ακόμα. Ο Ισαγγελεύς μου μας έδωσε επίσης και την ομιλία του, την οποία θα μοιράσουμε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν άλλον εμπειρογνώμονα, έναν Γάλλο εμπειρογνώμονα, τον Ζων Ζάκ Κολομπή, επικεφαλής της Μονάδας για τις Διεθνείς Σχέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, από το δικό του παρατηρητήριο. Και από τη δική του εμπειρία θα μας μιλήσει για τους τρόπους συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών θα ήθελα άλλος ιδιαίτερος αν μπορεί να μας εξηγήσει τι είδους πρόβλημα, προβλήματα επιχειρησιακά αντιμετωπίζετε όταν περνάτε από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό και μετά στο διεθνές επίπεδο. Θα υιοθετήσουμε την ίδια μέθοδο των συζητήσεων. Λοιπόν, σας δίνω πρώτα το λόγο. Pardon. J'imagine que ça fonctionne mieux. Με το μικρόφωνο είναι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να σας κάνω μια παρουσίαση σχετικά σύντομη. Σε μια πρώτη φάση και να έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Είμαι Γάλλος αστυνομικός, όπως είπε η Πρόεδρος, ε, από την δίωξη της Γαλλίας. Ε, για όλες τις αρχές επιβολής του νόμου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εγώ είμαι αρμόδιος για όλες τις διάβλους επικοινωνίας ε, ανάμεσα στις, ε, στα λειτουργικά και θεσμικά τμήματα των αστυνομικών αρχών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρω ότι λειτουργείται σε ιταλικό αστερισμό. Ε, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ όμως παρόλα αυτά κάποια πράγματα στην ε, Γαλλία δεν έχουμε τέτοια ε, φαινόμενα ε, μαφίας όπως στην Ιταλία. Υπάρχουν φυσικά οργανωμένες ομάδες που υπονομεύουν τη δράση του κράτους. Η απουσία της μαφίας στη Γαλλία δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν πάσχουμε από την οργανωμένη εγκληματικότητα. Ε, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι πολυσχηδής η οργανωμένη εγκληματικότητα στην Γαλλία και θα ήθελα να σας βοηθήσω ε, αναφερόμενο σε, σε κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Εσείς μιλήσατε για τη μαφία στην ε, Ιταλία. Βλέπουμε ότι μέσα στην αίθουσα είμαι ο μόνος ε, που ε, δεν είμαι Ιταλός και παρόλα αυτά εδώ και 7 χρόνια ε, ήμουνα στην αντίστοιχη υπηρεσία και είδα την κυρία Μπορσελίνο και θα ήθελα απλώς ποτινόμενος αυτή να της πω πόσο εκτίμησα που συνεργάστηκα με τον κύριο Φαλκόνο και τον αποθανόντα αδελφό της ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, στην Ιταλία. Μπορώ να σας μιλήσω ε, για την τουρκόφωνη και ρωσόφωνη μαφία στη Γαλλία ή για την λατινοαμερικανική, αμερικανική μαφία. Μπορώ να σας μιλήσω για τη νέα μόδα στην Ευρώπη, δυστυχώς, σας το πω έτσι, η περιοδεύουσα εγκληματικότητα από τις Χώρε ε, τη ε, Ανατολικής Ευρώπης. Όμω δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Θέλω να σας μιλήσω για τη γαλλική οργανωμένη εγκληματικότητα, αυτή δηλαδή που ουσιαστικά ε, διαπράτεται από εγκληματίες που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, δρούν στη Γαλλία ή με βάση τη Γαλλία προς την Αλοδαπή τι γίνεται λοιπόν με το, την γαλλική οργανωμένη εγκληματικότητα. Μπορέσαμε να προσδιορίσουμε και μια τυπολογία. Ξέρω ότι στις διεθνείς ε, οργανώσεις δεν μην ε, συζητούμε ε, και δεν επεκτηνόμαστε για αυτό το θέμα το, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Για μας όμως 75% της οργανωμένης εγκληματικότητας είναι γαλλικής υπηκότητας. και αυτό το 75% από το 75% ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προέρχεται από το εμπόριο κανάβεως ε, με ε, έδρα τα προάστια του Παρισιού. Πρόκειται για εγκληματικές ομάδες που γνωρίζουμε εδώ και καιρό διαρκούν ε, ε, και ε, συνεχίζουν τη δράση τους ΕΣΑΗ e, και μιλάμε για τη Λίλη, για την κατεβαίνοντας προς τα κάτω, φτάνοντας μέχρι την Κιανή ακτή, αυτή είναι η γραμμή δράσης αυτών των ομάδων και φτάνουμε φυσικά στην Κορσική. Τι εννοούμε τώρα μιλώντας για την Κορσική μαφία. Est-ce que c'est une mafia comme Cosa ε, λοιπόν, ε, η, Κορσική είναι, έχει 150.000 ε, κατοίκου. μιλάμε για εντελώ διαφορετικέ τάξει σε μεγέθους. Από το 2008 και μετά, όταν ξαναρχίσει στην Κορσική η επανασχεδίαση της εγκληματικής αρχιτεκτονικής ή η κίνηση των τεκτονικών πλακών της Μαφία στην Κορσική, σημειώθηκαν 67 ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μέχρι σήμερα. Οι ομάδες αυτές ε, παραδοσιακά είναι, σας είπα, από, στη γραμμή από την Κιανή Ακτή μέχρι το Παρίσι, τυχερά παιχνίδια, εκβιασμός, ένοπλη ληστεία, διαφθορά, ε, κερδοσκοπία στο ε, τομέα της ακίνητης περιουσίας. Έχουμε διακλαδώσεις στην Αφρική Λατινική Αμερική με τα καζίνο, τα ξενοδοχεία κτλ. Ε, οι ε, Κορσικανοί και οι Μασαλιέζοι συνεργάζονται μεταξύ τους ε, και αυτό συνεχίζεται εδώ και 30 χρόνια. Ε, οι ε, μασαλιώτες λοιπόν, ε, νονοί, συνεργάζονται με τους κοσικανούς νονούς και ασχολούνται με αυτά που σας είπα, τυχερά παιχνίδια, ξενοδοχεία, καζίνο, στη Νίκη στην Τουλό και στη Μοπελιέ έχουν επεκταθεί, κυρίως όταν έχουν περισσότερο προσωπικό, αλλιώς περιορίζονται στη Μασαλία. Στη Λίλη έχουμε επίσης συνεργασία με εγκληματικά στοιχεία από το Βέλγιο, στο, ε, στη Λιόν ε, έχουν αποσαρθωθεί διάφορα κυκλώματα ε, και φτάνω τώρα στα προάστια του Παρισιού όπου παρατηρείται η πιο έντονη οργανωμένη εγκληματικότητα. Γενικευμένο φαινόμενο, ειδικό στη Γαλλία και συνδέεται με τις μασικές εισαγωγές εδώ και χρόνια κανάβιος από το Μαρόκο μέσα από τη, μέσω της Ολλανδίας ή της Ισπανίας. Ο ο τζίρο ανέρχεται σε 3 δις ευρώ περίπου ε, το χρόνο και 250 τόνοι το χρόνο καταναλώνονται στην Γαλλία. Είναι η βασική πηγή παρανόμου εισοδήματο ε, στη Γαλλία και προ υπενθύμηση το εμπόριο ναρκωτικών των άλλων μεγάλων προϊόντων, ε, δηλαδή συνθετικά ναρκωτικά, κοκαίνη και η ηρωίνη, βάσει τη αρμόδια υπηρεσία ανέρχεται σε ένα δις μόνο η πλειοψηφία αυτών των ε, εγκληματικών ομάδων ε, που εμπλέκονται και στι εισαγωγέ ε, και στη μεταπόληση προέρχονται από αυτά τα προάστια, σα το είπα. Έχουν συνάφεια με του παραγωγού στο Μαρόκο και αυτό διευκολύνει τι συναλλαγέ και επίση τα προϊόντα επιστρέφουν στο Μαγκρέμπ ή σε διάφορε χώρε, είτε στο Μαρόκο, είτε στην Τινησία, είτε στην θα είμαι σύντομο γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Να σας πω πώ έχει η οργάνωση. Είναι σε τρία επίπεδα ε, η οργάνωση αυτών των ε, ομάδων περίπου σε 400 ε, ένοχες, ας το πούμε, πολυκατοικίες των προαστίων αντιπαλότητες ε, τώρα που υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορες, ε, στα διάφορα μέλη των εγκληματικών ομάδων και ανάμεσα σε εγκληματικές ομάδες για τον έλεγχο του ε, εδάφους είναι πάρα πολύ μεγάλες και νομίζω ότι ο Γενικός Αγγελέας θα καταλάβει ε, περί τίνος πρόκειται. υπάρχει χρήση όπλων και διάπραξη άλλων εγκλημάτων. Οι χοντρέμποροι ε, προωθούν εκατοντάδες κιλά καναβέως έχοντας άμεση σχέση, όπως σα είπα, με τους παραγωγούς, γιατί πρέπει να προπληρώσουν το εμπόρευμα και στη συνέχεια πρέπει να μετακινηθούν γρήγορα στην Ολλανδία ή στην Ισπανία για να ε, παραλάβουν τα φορτία. Ε, στη συνέχεια, πέρα από την κάναβη, έχουμε και την απειλή άλλων προϊόντων και προσοχή, διότι το εμπόριο τη ε, κοκαίνη έχει αυξηθεί ανησυχητικά και ξέρουμε ότι αποθηκεύεται η κοκαίνη και προωθείται από την Δυτική Αφρική. Αυτές οι εγκληματικές ομάδες εισάγουν λοιπόν ε, κοκαίνη στην Γαλλία και μεταφέρουν την ε, κοκαίνη που εκδημοκρατίζουν έτσι, μέχρι ε, τα προάστια, μέχρι τα, τις σκάλες των πολυκατοικιών αυτών σε αυτές τις επίμαχες συνοικίες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα του εμπορίου ναρκωτικών. η αστική που τώρα έχει γίνει περιαστική η εγκληματικότητα αγγίζει πλέον και τη Γαλλική ύπεθρο. Ε, πάνω πάνω στην πυραμίδα, τη, ε, της, πάνω πάνω στην εγκληματική πυραμίδα, έχουμε ε, κάποιες, ε, κάποιες τέτοιες συνοικίες ε, που έχουν ανέβει στην κορυφή αν θέλετε αυτών των συνοικιών. Είναι αυτοί οι χοντρέμποροι που εισάγουν σε κάθε φορτίο τόνους κανάβιους και είναι πολύ καλά διαρθρωμένες αυτές οι ομάδες, κατέχουν τον τρόπο συναλλαγής, διαφθείρουν υπαλλήλους των αστυνομικών αρχών της Ολλανδίας και της Ισπανίας που αποφελούνται από αυτό και κάνουν κάνουν επενδύσεις στη Γαλλία αλλά κυρίω ε, στην Αλοδαπή. Οι υπεύθυνοι, και θα δείτε στη συνέχεια γιατί επιμένω για αυτό, ε, βρίσκονται κατεστημένοι στο, στη Νότια Ισπανία, στην ε, Ολλανδία ή στι Μαροκινέ ακτές. Ε, το διακύβευμα από οικονομική πλευρά είναι τεράστιο, εξυπακούεται αυτό και ε, πέραν αυτού υπάρχουν και συναφεί ε, εγκληματικέ πράξει. Σήμερα στη Γαλλία θεωρούμε ότι 70 80% των 50 ξεκαθαρίσματων λογαριασμών που σημειώνονται στη Γαλλία σχετίζονται με την εκαναβή προβλήματα με την ποιότητα του προϊόντος, την ποσότητα ποιότητα του προϊόντος, ε, το μη σεβασμό κάποιων κανόνων σε σχέση με τη μεταφορά και τον έλεγχο κυρίως ε, του, της του τους ε, σε εισαγωγικά. ζητούν λοιπόν λίτρα είτε στη Γαλλία είτε στην Αλλοδαπή για να εκβιάσουν κάποιου, κλέβουν εμπορεύματα γιατί κάποιε ομάδες ειδικεύονται σε ένοπλες ληστείες των διακινητών για τους οποίους σας μιλούσα ή κατά των εισαγωγέων για τους οποίους σας μιλούσα προηγουμένω. 7,5 λεπτά. Ιδού, ε, νομίζω ότι σας εξήγησα ε, ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα αυτού του φαινομένου. Α, και στη Γαλλία θέλω να σας πω κάτι. Όχι ε, για να μετατοπίσω την εστίαση της συζήτησή σας, αλλά διότι είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα πώς χρησιμοποιούμε στη χώρα μας ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Όλα περιστρέφονται γύρω από τη διεθνή συνεργασία. Αυτό νομίζω το έχετε πλέον αντιληφθεί. Ε, θέλουμε να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση, μια ε, ε, έχουμε και εμείς προσδιορίσει μία αρχιτεκτονική. Δηλαδή για την διεθνή αστυνομική συνεργασία ε, από το 2000 και μετά η Γαλλία θέσπισε ένα ενιαίο σημείο εισόδου ως προς την κεντρική διεύθυνση της δίωξής μας ενώνοντας όλα τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν οι ερευνητές μας Αντερπόλ, Europol, Schengen, γιατί ε, έχει θεσμοθετηθεί λοιπόν η συνεργασία και έχει εισέλθει στα πλαίσια της ποινική ε, δίωξης. Ε, θα μου πείτε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε στην Ευρώπη. Συμβαίνει αυτό και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσε. Η ιδιαιτερότητα της γαλλικής, αυτού του γαλλικού τρόπου συνεργασίας, αυτής της γαλλικής αρχιτεκτονικής είναι ε, η εξή ε, τελωνιακή, δικαστική, αστυνομική ε, και τα λοιπά συνεργάζονται επί 24 ώρου βάσεως, δηλαδή όταν υποβάλλεται αίτημα από αλλοδαπούς εταίρους είναι διαθέσιμοι πάλι ούτως ώστε να διεκπαιρεώσουν καθήκοντα που σχετίζονται με την αστυνομική συνεργασία. Παραδείγματο χάρη, επιγόντω ένα ε, δικαστή από τη Λιθουανία ή από την Ισπανία εκδίδει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Έχουμε ενδείξει ε, για το που βρίσκεται ο φυγόδικο στη Γαλλία και σε πραγματικό χρόνο και 24 ώρε το 24 ολόκληρο το χρόνο έχουμε την έγκριση τη αστυνομία και μπορούμε να προβούμε στην ε, σύλληψη. Θα μου πείτε... Εντάξει, αλλά τι γίνεται με τα υπόλοιπα μέσα που έχετε ε, στην ε, διάθεσή σας. Ε? Σας είπα ότι θέλουμε να είναι συνεκτική η δράση μας και κυρίως ολιστική. Υπάρχουν, πέρα από αυτά τα εργαλεία που σας περιέγραψα, τα διμερή εργαλεία. Ας πάρουμε το εμπόριο ναρκωτικών, παραδείγματο χάρη. Ας πάρουμε, εφόσον σας μιλούσα για την Δυτική Αφρική και για το δρόμο που από το Μαρόκο προς την Ισπανία, όχι για κάποιο λόγο, αλλά επειδή είναι πολύ χαρακτηριστική Ξέρουμε ότι φτάνει από τη Λατινική Αμερική η κοκαίνη στην ε, Δυτική Αφρική. Ξέρουμε ποιε χώρε παράγουν, είναι τρει. Ε, ξέρουμε ποια είναι τα κράτη ε, που μεταφέρουν, αν θέλετε, και είναι τα αεροπλανοφόρα των χωρών παραγωγών. Ποια μέσα χρησιμοποιούμε, λοιπόν, ούτω ώστε να είναι συντονισμένη η καταστολή σε σχέση με τη δράση των εταίρων μα. Έχουμε φυσικά αξιωματικού σύνδεση και δεν τονίζουμε παρκώ το ρόλο του. Αυτή η αξιωματική σύνδεση ε, ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, ε, σε πάνω από 90 ε, χώρες ε, έχουμε τέτοιους αξιωματικούς και έχουν αρμοδιότητες 146 χώρες. Στη Λατινική Αμερική ασχολούνται με τη κοκαίνη, στη Βενεζουέλα, στο Περού, στη Βραζιλία. Παντού έχουμε τέτοιους αξιωματικούς. Φυσικά όπως και άλλοι είμαστε σε διαρκή επαφή με την Αμερικανική αρμόδια αρχή για να ξέρουμε τι γίνεται στην Καραϊβική για το περίφημο GATF στην για να είμαστε στην γαλλική επικράτεια αλλά ε, ε, εγκύτερα στις ε, ζώνες παραγωγής. Έχουμε από την Κεντρική Υπηρεσία Δίωξη των Ναρκωτικών επιτόπου μία μονάδα ούτως ώστε να δράσουμε προτού φύγει από τη χώρα αυτή το εμπόρευμα και εκεί συνεργαζόμαστε με την Αγγλία, την Ιταλία, την Γερμανία για τους ίδιους λόγους. Φυσικά χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες μέσα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ για τις πλατφόρμες σύλληψη των ε, σκαφών που διέρχονται τον ε, διαπλέον τον Ατλαντικό. Ε, έχουμε επίσης τους αξιωματικούς μας στην Δυτική Αφρική, στον Τακάρ παραδείγματος χάρη, και στην Γκάνα, στην Άκρα, όπου έχουμε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και πάλι τους Ολλανδούς, τους Ισπανούς, τους Ιταλούς, Πορτογάλους, τους Γάλλους, να εννοείται, τους Βρετανούς. Και στη συνέχεια έχουμε πολλοί αριθμούς τέτοιους αξιωματικούς στο Μαρόκο και στην Ισπανία για να επανέλθω στο εμπόριο ε, ε, που σχολίαζα νωρίτερα, θα σας έλεγα ότι η Γαλλία πιστεύει ότι Πέρα από αυτά τα εργαλεία διεθνού συνεργασία, ε, όπω η Europol, και αν θέλετε μπορώ να επανέλθω συνέχεια σε αυτό, πέρα από αυτό υπάρχουν διάφορε επιχειρήσει ε, που μπορούν να ε, διεξαχθούν μόνο σε πλήρη συνεργασία και συγχώνευση όλων των εταίρων, τη δράση των εταίρων. Γι' αυτό στην Μαδρίτη, στη Μάλαγα, στην Βαρκελόνη, έχουμε στο Αλικάντη, σε διάφορα μέρη της Ισπανίας έχουμε επιτόπου ε, μονάδες ε, και επίσης ε, ε, Στην Νότια Ισπανία, η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε ένα κοινό αστυνομικό τμήμα ε, που και θα μπορούσαμε εμείς να αποσπάσουμε αξιωματικούς ε, σε αυτό το αστυνομικό τμήμα ε, στην Αλζεσίρα, στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο. Αυτό φυσικά υπό την επιφύλαξη άλλων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά όπως σας έλεγα και προηγουμένως και για να προχωρήσω λίγο περισσότερο τη σκέψη μου, οι δύο κυβερνήσει τον Απρίλιο του 2010 υπέγραψαν μια συμφωνία, Υπουργοί Εσωτερικών συγκεκριμένα, για να δημιουργήσουν μόνιμε μονάδε πληροφοριών στη Γαλλία για την ε, καταστολή του λαθρεμπορίου και την εξάρθρωση ε, των συμμοριών ε, in situ δρούμε, δηλαδή εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι έδρες αυτών των οργανωμένων ομάδων, συγκεκριμένα στην Νότια Ισπανία. Ε, επεξεργάζονται πληροφορίες ε, λοιπόν σε αυτή τη μονάδα, πληροφορίες που συλλέγονται από όλους αυτούς τους αξιωματικούς ε, στη συνέχεια όσοι ειδικεύονται στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και στο ξέπλυμα χρημάτων στο ίδιο τμήμα και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ισπανικές αρχές καταλήγουν σε, στα συγκεκριμένα στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία των εγκληματικών ομάδων που βρίσκονται εκεί πέρα το 2010 θα σας δώσω τα αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων. 18 τόνους ε, κανάβεως, 600 ε, κιλά κοκαίνης, 80 οχήματα, 1.600.000 κατασχέθηκαν, 174 ε, εγκληματίες παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη, εκ των οποίων 150 ήταν εντελώς άγνωστοι στις γαλλικές αστυνομικές υπηρεσίες. Έχουμε φτάσει στα 15 λεπτά. Quelques instants Άλλο λίγο ακόμη, έχω να σας πω κάποια άλλα. Ε, είπαμε υπό την επιφύλαξη των μέσων διεθνού συνεργασία. Ποια είναι η γαλλική θέση λοιπόν γι' αυτό, η, Γαλλία επιθυμεί να ε, αξιοποιήσει στο έπακρον τη συνεργασία με την Europol, διότι πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητά τη, γνωρίζουμε ε, την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων τη έρευνα που γίνεται στην, ε, στον οργανισμό αυτών και Πιστεύουμε ότι ε, ήταν πολύ αποτελεσματική η καινοτόμως πρωτοβουλία που άρχισε πέρυσι στις αρχές του έτους, ε, δηλαδή ε, πέρα από την, δικαστική, την στρατιωτική αστυνομία, την ε, αστυνομία και τα γαλλικά τελωνία, ε, προβλέψαμε το ενδεχόμενο συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές ε, τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τους Europol. Η συνεργασία περνάει μέσα από την κεντρική υπηρεσία που διευθύνω εγώ. Εντάξει, ξέρω ότι έχουμε την τάση να επιλέγουμε διαρκώς την κεντρική διαχείριση. Στη Γαλλία μας αρέσει αυτό γιατί είμαστε φιλοβασιλικοί ως γνωστόν, αλλά θέλω να πω ότι ε, χρειάζεται αυτή η κεντρική διαχείριση για να μπορέσουμε να συντονίσουμε την δράση όλων αυτών των υπηρεσιών. Έτσι καταφέρνουμε συστηματικά να χρησιμοποιούμε τα αρχεία της Europol επί τη βάση των δεδομένων που συλλέγουν τα κράτη-μέλη. Στο στάδιο που, βρίσκεται τώρα η, λειτουργία της Europol αλλά και σε σχέση με τη λειτουργία των αστυνομικών αρχών αλλά και την φιλοσοφία που ακολουθούν οι δικαστικοί λειτουργοί στη Γαλλία προκρίνουμε ε, αυτόν η χρήση των στοιχείων των βάσεων δεδομένων της Europol η οποία όμως δεν πρέπει να καταστεί υποχρεωτική γιατί θα γίνει αντιπαραγωγική. Πάλι σε σχέση με την Europol είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την επιτυχία ε, των ευρωπαϊκών εργαλείων πριν τρεις πυλώνες ε, καλά Σέγγεν ε, είναι η καθημερινή αστυνομική συνεργασία δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ σε αυτό για πάρα πολλά ζητήματα αλλά πιστεύω και θα κλείσω εδώ αν συμφωνείτε κι εσείς que l'utilisation de ces outils η χρήση αυτών των εργαλείων σε μια, ένα παγκοσμιοποιημένο τοπίο ε, και το ίδιο ισχύει και για τις εγκληματικές πράξεις, απαιτεί μια εξισορροπημένη χρήση των ευρωπαϊκών μέσεων καθώς και των μέσων της Ιντερπόλ. Σας υπενθυμίζω ότι η Interpol, ε, στην Ιντερπόλ συνεργάζονται 180 διαφορετικοί κράτη και προσφέρονται πάρα πολλέ δυνατότητε συνεργασία. Θα πρέπει τώρα, στην περίπτωση ηλιτότητα, να αποφύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη, οποιαδήποτε απώλεια δυναμικού και ενέργεια. Ε, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο Evergreen και ε, την Interpol και την Europol. Και έχουμε εδώ του ναι. διευθυντέ των δύο οργανισμών. Δηλαδή, χρειάζεται συνεργατική σχέση και γι' αυτό στη Europol θέλουμε να εγκαταστήσουμε την πλατφόρμα για το κυβερνοέγκλημα και θα υποστηρίξουμε την εγκατάσταση Σιγκαπούρη ενό μέσου αντίστοιχου ε, από πλευρά της Ίντερπολ. Όμω χρειάζεται συνεργασία, πρέπει να βρούμε του τρόπου για να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η θέση της ε, Γαλλίας. Ε, αυτό είπαμε και στο... Διευθυντικό Συμβούλιο και των δύο οργανισμών όταν κληθήκαμε να τοποθετηθούμε. Δεν θέλω να επαναλάβω εξάλλου, δεν θα το προσπαθούσα κάνε ε, αυτά που είπε ο εισαγγελέα Αγκράσο. Ε, θα μπορούσα να μιλήσω λίγο για τις μελλοντικέ ε, προκλήσεις και για αυτό που εμείς στην δίωξη της γαλλία ή στο δικαστικό σώμα της Γαλλία μπορούμε να περιμένουμε από εσάς και από την εμπειρία σας. Ο εισαγγελέα Γκράζο μα μίλησε προηγουμένω για την οδηγία για την διατήρηση και αποθήκευση των στοιχείων. Πλήρω θα συμφωνήσω μαζί σας και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που ε, προκύπτει δυστυχώς από την πρόσφατη εγκληματική επικαιρότητα της Γαλλίας. Ε, όλοι είδαν τι έγινε στην ε, Τουλούζη. Στο Μοντοπά δεν είναι μόνο τα πραγματικά περιστατικά, αλλά για την ανάγκη και το ενδιαφέρον ε, των διοκτικών αρχών και τι αντιμετώπισαν οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Ταυτοποιήθηκε ε, αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή του δράματος και η δίωξη ε, και η έρευνα θα δείξει πώς κατάφερε να στήσει ε, μια τέτοια τρομοκρατία. Διαπιστώσαμε ότι είχε πάει στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν. Σε μια τέτοια έρευνα είναι προφανές ότι αυτό ε, γίνεται ε, αναδρομικά. Είναι μια έρευνα που γίνεται στο παρελθόν, προς τα πίσω. Και τα φαινόμενα που έχουν σημασία για την έρευνα μπορεί να ανάγονται σε περισσότερα έτη. Ε, στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι χρειάζεται να προστατεύονται οι ατομικές ελευθερίες του καθενός μας, αλλά ταυτόχρονα φοβόμαστε πάρα πολύ ότι αν μειωθεί ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων μπορεί να είναι εις βάρος τέτοιων ερευνών. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να πω, αυτός ο νεαρός πήγε στην Ισλαμαμπάτ και δεν μπόρεσε να πάει από το Παρίσι γιατί δεν υπάρχει επευθείας πτήση αναγκαστικά χρησιμοποίησε ενδοκινοτικές πτήσεις. Και πολύ σύντομα ε, επανέρχομαι στο θέμα PNR της ε, λίστας των στοιχείων επιβατών. Και εκεί ακόμα, αν δεν συμπεριληφθούν οι ενδοκινοτικές πτήσεις σε αυτό τον κανόνα του PNR, γίνεται αδύνατη κάθε είδους έρευνα. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε για να επανέλθω στην οδηγία για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων. Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι βουλευτές και για τη χρήση που θα πρέπει να κάνουμε των μέσων της Ιντερπόλ που συνεισφέρουν όλες μας οι χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της χρηματοδοτικής πτυχής. Σας παρακαλώ μην παραλείψετε στην οδηγία αυτή να προβλέψετε ανταλλαγή πληροφοριών με ε, τους διεθνείς οργανισμούς γιατί στην παρούσα οδηγία και στο κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει ένα μικρό νομικό κενό. Δεν αναφέρεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τους διεθνείς θεσμούς και αυτό μας δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Αυτά, Πρόεδρε, θα είχα σίγουρα πολλά και άλλα να πω, αλλά δεν θα είχαμε χρόνο για τις ερωτήσεις. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Σας ευχαριστώ, κύριε Κολομπή. Εμείς έχουμε χρονικά προβλήματα και έχουμε δαμόκλειο σπάθη από πάνω μας. Θα παρακαλέσω τη γραμματεία να δώσει στον κύριο Κορκοράνα μέσα στο λόγο να ξεκινήσει μετά ο γύρος των ερωτήσεων. Ο κ. Κορκοράν είναι υπεύθυνο υπηρεσία για τα... τι Ιρλανδίε. Ο κ. Κορκοράν. και θα μιλήσει για το κόψιμο, δηλαδή τι γίνεται όσον αφορά τον εντοπισμό κατά σχέση των προϊόντων εγκλήματος. Γνωρίζουμε η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών συζητά το θέμα αυτό, την οδηγία για τις κατασχέσεις, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έκανε πρόταση για έναν κανονισμό όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των εντολών κατάσχεσης. Ζητώ από τον κύριο Κόρκοραν να μας πει ποια είναι η εμπειρία του όσον αφορά τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισε καθημερινά σαν επικεφαλής υπηρεσίας προϊόντων εγκλήματος Ιρλανδίας και για τα προβλήματα αυτά που δεν γνωρίζουν ε, σύνορα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας. Ε, είμαι επικεφαλής ε, διευθυντής ε, του Γραφείου Κατασχεθέντων Προϊόντων Εγκλήματος της Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα σας δώσω γενικά μία παρουσίαση της υπηρεσίας μας Επίσης, να σας πω και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος και ε, σχετικά ζητήματα. Και θα αφιερώσω ε, πολύ λίγο χρόνο ε, στις εξελίξεις των τελευταίων 15 ετών που υπάρχει η υπηρεσία μας και πώς αλλάζουν οι τάσεις ή πώς άλλαξαν καθόλου αυτή τη 15 ετία. Για να καταλάβουμε τις εξελίξεις ε, ε, της ε, κατάστασης, κατάσχεσης που δεν συνδέεται με καταδίκη, θα πρέπει λίγο να σας εξηγήσω τι συνέβαινε πριν το 1994. με ένα νόμο του 1994 που αφορούσε την κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος. Ήταν πάρα πολύ σημαντική τότε η νομοθεσία και πολλές οι αλλαγές στο νόμο αλλά χρειαζόταν πρώτερη καταδίκη για να δοθεί ένα ένταλμα κατάσχεσης. Ε, είχε σχέση με την απαγγελία συγκεκριμένης κατηγορίας και την καταδίκη του προσώπου για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προβούμε σε κατάσχεση των διαφόρων ε, προϊόντων εγκλήματος ε, και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και λοιπά. παρά τις σημαντικές εξελίξεις που είχαμε στη συνέχεια ε, στο ποινικό δίκαιο παρέμειναν ε, κάποιοι σοβαροί εγκληματίες που ε, είχαν τη δυνατότητα να απακιστρώνονται από την εγκληματική πράξη οι ίδιοι επιχειρησιακά ή μέσω ενός περίπλοκου χρηματοοικονομικού συστήματος να διαφεύγουν. Το 1990, στα μέσα της δεκαετίας, είχαμε πολλές τέτοιες ε, οργανωμένες ε, εγκληματικές οργανώσεις που ε, κατάφεραν να εκφεύγουν των ποινικών δικαστηρίων. Και τελικός καταλήτης για τη δημιουργία της υπηρεσίας μας ήταν δύο δολοφονίες το καλοκαίρι του 1996 ενός δημοσιογράφου και ενός ε, ε, αστυνομικού. Και το ε, αποτέλεσμα αυτών των τραγικών γεγονότων ήταν η νέα νομοθεσία. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για την Επιτροπή σας. Απλώς θέλω να σας πω να σας αναφέρω μία παράθεση ενός εξέρχοντος δικαστικού τότε που ερμήνευσε τον νόμο. Και ε, η ουσία ήταν ότι αυτό έγινε λόγω ανάγκης, αλλά ε, και για να υπάρχει μια στενή επιτήρηση από τα δικαστήρια. Αντίστοιχα, ε, συμβαίνουν και με ένα νόμο που προέκυψε από την αρχή της αναλογικότητας και της εξισορρόψης δικαιωμάτων μεταξύ του ε, λόγω ατόμου και γενικότερα της κοινωνίας. Έρχομαι τώρα στην υπηρεσία μας αυτή καθ' αυτή. Είναι μικρή σε μέγεθος ε, ε, σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα και ισχύοντα. 70 είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που είναι μικρός αριθμός σε σχέση με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα. Και έχουμε ε, στελέχωση από διάφορα υπουργεία. Όπως βλέπετε εδώ, η μισή, 36, είναι αστυνομική, 12 ε, ε, είναι εφοριακή, 5 είναι από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προστασίας. Επιπλέον, έχουμε ένα νομικό υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, πέντε αναλυτές και συνολικά 11 διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους. Όπως σας είπα, η υπηρεσία μας είναι πολύ μικρή ως προς το μέγεθος σε σχέση με τις ε, διεθνείς οργανώσεις. Και αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος του πληθυσμού και της αστυνομίας. Η αστυνομία μας αριθμεί 14.000 ε, ε, περίπου στελέχη, αλλά η αποτελεσματικότητά μας είναι προφανής, παρά το μικρό μας μέγεθος. Ε, οι στόχοι της υπηρεσίας αυτής καθ' αυτής, που από την νομοθεσία, ε, αναφέρονται απλά ε, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ε, εντοπίζουμε τα προϊόντα εγκλήματος ή τα φερόμενα προϊόντα εγκλήματος και να προβαίνουμε στις ε, διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο, να κάνουμε οποιασδήποτε έρευνες χρειάζονται για το σκοπό αυτό. Είναι γενικός ορισμός, ας πούμε, της αποστολής μας και πάρα πολύ γενική στόχη και με πολύ απλό τρόπο σας τους αναφέρω. Η υπηρεσία αυτή καθ' αυτή περιγράφεται ως διεπιστημονική διακλαδική υπηρεσία, ε, διακλαδική μάλλον. Έχουμε ε, αστυνομικούς, εφοριακούς, ε, υπαλλήλους των κοινωνικών υπηρεσιών που συνεργάζονται και μοιράζονται πληροφορίες με ένα κοινό στόχο. Οι ερευνητικέ δραστηριότητε υποστηρίζονται από λογιστέ, δικηγόρου, εμπειρογνώμονε, δικού μα υπαλλήλου, που έχουν όλοι την εξουσία να ερευνούν και να ανακρίνουν και να προβαίνουν και ε, σε οποιαδήποτε ε, κατάλληλη ενέργεια. Εδώ σας αναφέρω τις διάφορες υπηρεσίες που απαρτίζουν ε, το γραφείο μας και πάλι επειδή είναι σύντομο ο χρόνος δεν θα επεκταθώ σε κάθε μία ξεχωριστά. Θα ήθελα μόνο να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. Πρόσφατα η υπηρεσία μας επικεντρώθηκε περισσότερο στην ανάλυση ε, και στην προετοιμασία υποθέσεων για τα δικαστήρια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ευεργετικό. Δηλαδή, όλη η πληροφορία και τα στοιχεία που συλλέξαμε, που συλλέγαμε μάλλον στο παρελθόν, τα αγνοούσαν και προτιμούσαν με πιο ε, άμεσα πιστήρια. Ενώ πρόσφατα αναλύουμε τον τρόπο ζωής, το εισόδημα και άλλα στοιχεία ε, των εγκληματιών για να ε, έχουμε μια εικόνα το πώς έχουν φτάσει ε, σε αυτό το προϊόν του εγκλήματος. Ε, έχουμε διάφορες ικανότητες, δεξιότητες και οι υπάλληλοι μας συνεργάζονται σε ομάδες υπό την ίδια στέγη, υπό τον ίδιο προϊστάμενο υπάλληλο που είναι συνήθως αστυνομικός και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην αρχή της ισότητας μεταξύ των διαφόρων ε, μονάδων και υπηρεσιών που συνεργάζονται. Δηλαδή ε, συνεισφέρουν όλοι ανάλογα και εξίσου και ε, είναι πάρα πολύ αξιόλογο το έργο όλων των εργαζομένων. Η νομοθεσία που καλύπτει τη λειτουργία της υπηρεσίας ε, ορίζει πώς μπορούμε να βρούμε στοιχεία στις έρευνες, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο όλων ε, για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας είναι η εξουσία που έχουν και η δυνατότητα οι υπόλοιποι ε, υπάλληλοι εκτός των αστυνομικών να δρουν ανώνυμα και να έχουν προστασία από τον κανονισμό υπηρεσιακής τους κατάστασης ως προς την ανωνυμία. Θα πρέπει και αυτό να υποθεί. Η υπηρεσία λειτουργεί με τρόπο πάρα πολύ εστιασμένο κάθε φορά και στρέφεται κατά προσώπων. Δεν έχουμε μια γενική παρακολούθηση, έρευνα. Επιλέγονται πάρα πολύ ε, προσεκτικά οι υπαλλήλοι μας γιατί χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ε, και ε, δεξιότητες ε, σε σχέση με τα εγκλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Σας είπα ότι είναι διακλαδική η δουλειά μας από πολλά υπουργεία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην πράξη. Και σε μεγάλο βαθμό, χάρη σε αυτό, έχουμε και τις επιτυχίες που γνωρίζουμε σήμερα. Δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας της πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών μας ε, είναι ε, πραγματικά ε, λύση των παραδοσιακών ε, δυσκολιών που γνωρίζουν όλες οι μεγάλες γραφειοκρατικές δομές. Κάθε στόχος έχει μια επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί με τρόπο συντεταγμένο και συγκεντρώνει στοιχεία. Έχουμε μια ειδική στρατηγική για να αποκαλύπτουμε τα προϊόντα κλίματος και συνεργάζονται πάρα πολύ καλά όλες οι υπηρεσίες ε, του γραφείου μας. Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία μας είναι ένας νόμος του 1996. Δεν προτείνω σε καμία περίπτωση να αναφερθώ στις ε, λεπτομέρειες. Τα βασικά χαρακτηριστικά του νόμου είναι ε, ότι υπάρχει κατάσχεση αστικού δικαίου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη ποινική καταδίκη. Τα τελευταία χρόνια ε, έχουν προσβληθεί αυτά και ε, έχουν φτάσει μέχρι το ανώτατο δικαστήριο. Ε, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για νομική συνδρομή και προστασία και ε, κάλυψη των εξόδων καλή τυπή στην Πόνα Φίντε. Για μια επταετή περίοδο που μεσολαβεί από την έκδοση του εντάλματος κατάσχεσης μέχρι την πραγματική δίμευση ή αξιοποίηση ε, του περιουσιακού στοιχείου. Οι εξουσίες που συνδέονται ε, από με την εφορία και τις κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να ε, χρησιμοποιούνται από κοινού ή ξεχωριστά. Πάντως όλες οι εξουσίες και όλες οι αρμοδιότητες ε, φροντίζουμε να ε, υλοποιούνται με τρόπο συντονισμένο. Έρχομαι σύντομα στη διεθνή διάσταση της εργασίας μας. Έχω φτιάξει μια διαφάνεια που δείχνει την κυριότερη διεθνή συνεργασία που έχουμε. Ε, δεν θα σας εκπλήξει ότι η περισσότερη συνεργασία μας και διάδραση γίνεται με συναδέλφους ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας και της αστυνομίας, αλλά ε, και πιο συχνά συνεργαζόμαστε και με τους Ευρωπαίους συναδέλφους και διεθνώς. Υπάρχει σήμερα ένα άτυπο δίκτυο υπηρεσιών κατάσχεσης προϊόντων εγκλήματος και είναι Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του 2007, πάρα πολύ χρήσιμη για μας στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών. Προσπαθώ να τηρήσω το χρόνο που μου δώσατε. Θα σας πω σε διεθνές επίπεδο ε, ποια είναι τα ζητήματα γιατί, ε, και ποιες οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και μπορεί να σας ενδιαφέρουν από καιρού καιρών ε, ε, βλέπουμε ότι άλλες ε, δικαιοδοσίες ανησυχούν κάπως για την ανταλλαγή προφοριών σε ό,τι αφορά τις έρευνες αστικού περιεχομένου, όχι ποινικού δικαίου και μετά από καταδίκη. Είναι ένα θέμα αναγνώρισης και επιβολής ενταλμάτων. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχουμε τελικά ε, διατίθενται ε, με έναν τρόπο που υπόκειται σε έλεγχο υψηλού δικαστηρίου και εποπτεία. Και επίσης ε, η αναγνώριση και επιβολή ενταλμάτων αστικού δικαίου είναι κάτι που δεν αναγνωρίζουν πολλοί, αλλά στη δική μας δικαιοδοσία ισχύει και υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά διεθνώς χρειάζεται ενδεχομένω μεγαλύτερη μελέτη. Η, Επίσης, ε, από κοινού, όταν κατάσχουμε ε, περιοσιακά στοιχεία με άλλες δικαιοδοσίες, υπάρχει ένα ζήτημα καταμερισμού εκεί. Ε, είναι κάτι που οδηγεί σε δυσκολίες από καιρό καιρό και αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα ερμηνείας των διεθνών μέσων και αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί ε, να οδηγήσει σε διαμάχες και διενέξεις. Ε, η υπηρεσία μας ε, λειτουργεί και φιλοδοξεί να είναι ένα μοντέλο για βέλτιστες πρακτικές. Έχει σημειώσει επιτυχίες στην Ιρλανδική δικαιοδοσία και παραμένει καθήκον μας να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο και αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόρκοραν που τα μας παρουσιάσατε όλα αυτά. Δίνω μέσω το λόγο στους συναδέλφους, συντονιστές και βουλευτές. Παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας. Αλλιώς θα αναγκαστώ να αφαιρέσω το λόγο γιατί φορετικά θα τελειώσουμε εγκαίρως. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ε, με τον κύριο, την κυρία Ματία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Μας ε, καθησυχάζετε, γιατί νομίζαμε ότι η μαφία ήταν μόνο στην Ιταλία. Επιτέλους, κύριε Κολομπή, μας είπατε ότι έχουμε και εμείς δική μας οργανωμένη εγκληματικότητα στη Γαλλία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην Ιταλία δεν ε, ε, ε, επικοινωνούμε όπως στην Ιταλία, μεταξύ, δηλαδή οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους σε σχέση με την κατάσχεση ναρκωτικών, για το ξέπλυμα χρήματος, για όλες αυτές τις επιτυχημένες επιχειρήσεις που μας περιγράψατε. Ε, επίσης υπάρχει έλλειψη συνεργασίας και με τους δημοσιογράφους, ε, οπότε το, το, το, κοινό, οι πολίτες ε, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει ακριβώς, αποσιωπούνται όλα, είναι κρίμα. Τέλος πάντων η γαλλική στρατηγική φαίνεται. Κατάλαβα τι επιδιώκετε, δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω τίποτα, θέλετε να αποθηκεύετε τα στοιχεία, δηλαδή η, έκθεση, η σχετική έκθεση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠ και το PNR. Ε, για τον ε, κύριο Κορκόραν θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλες τις δράσεις που έχετε αναλάβει στην υπηρεσία σας. Είναι πάρα πολύ θετικές, κυρίως για την κατάσχεση των προϊόντων εγκληματικών πράξεων. Σίγουρα θα υποφεληθούν πολλά κράτη από την εμπειρία. Σας ευχαριστούμε για ένα λεπτό. φαγιό. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, ήταν χρήσιμα αυτά που ακούσαμε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να στραφώ εν συντομία προς το εμπόριο ναρκωτικών στη Γαλλία. Έχω μια ερώτηση, όχι τόσο όσον αφορά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά το εμπόριο ανθρώπων, το δουλεμπόριο. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια στατηγική με 40 διατάξεις συγκεκριμένε για την καταπολέμηση του δουλεμπορίου. Ε, το έχετε σημειώσει αυτό, το έχετε παρατηρήσει. Στους εθνικούς ποινικού κώδικες που προσπαθούν να καλύψουν το εμπόριο λευκής σαρκός και την ε, δημιουργία μονάδων ερευνών, κοινών μονάδων ερευνών στην Ευρώπη για το δυσυνοριακό εμπόριο ανθρώπων. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, θα να ξέρω. Ε, μια πρωτοβουλία όπως Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών διότι ακούσαμε να μιλάμε και να με θέσετε σε αυτό το θέμα. Για την Άλντε, ο κύριος Νιούτον Ντόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τον κύριο Κολόμπη, έχω ένα ερώτημα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα βοηθούσε να έχουμε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα, ένα FBI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρώσεις ευρωπαϊκές για τους Εγκληματίε και φυλακές Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Ναι ή όχι μπορείτε να απαντήσετε αυτά. Είναι απλώ ε, σαν ένα Προ κατάλογος. Προς σαν ένα άδελφο. Πολύ ενδιαφέροντα. Τι γίνεται αν βρείτε ότι αυτοί οι κακοί έχουν περιουσία στην Ιρλανδία αλλά και στην Ελβετία ή στι ΗΠΑ Πώ Πώς συνεργάζεστε, ε, πώς μπορείτε να το κρατήσετε μυστικό σαν πράξη, σαν κίνηση, αλλά να πείτε στου Αμερικανούς και Ελβετού να βοηθήσουν και να το ψάξουν. Ευχαριστώ του Πρασίνου, Ο, Στά, ο κ. ECR, ο κύριος Κυρκόπ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που μπορεί να αφορά και τους δύο κυρίους, ίσως περισσότερο τον Ιρλανδό συνάδελφο. Οι επαφές, οι σχέσεις μεταξύ του έργου που κάνουν εκείνοι και τα, το Εθνικό Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά την οικονομική πτυχή του εγκλήματος είναι πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή και βάσει αυτών που συμβαίνουν τώρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα, όχι μόνο με το ξέπλυμα χρήματο, αλλά πιο συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται υποθέσεις διαφθοράς και το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Όλα αυτά γίνονται όλο και περισσότερο κοινές, κοινή προσπαθία των δυνάμεων της τάξεως και των εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό περισσότερο. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ ένα λεπτό ο κύριος Σόντεργαρντ. Δεν είναι εδώ. Προχωράμε. Ένα λεπτό ο εισηγητής ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα και τους δύο. Και τον κύριο Κολομπή και τον κύριο Κορκόρεν. Και είδαμε πόσο σημαντικά μοντέλα υπάρχουν και αλλού, εκτός Ιταλίας αποτελεσματικά μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα κατά πολέμηση οργανωμένου εγκλήματος. Και για τους δύο έχω το ίδιο ερώτημα. Τι μέσο, τι εργαλείο, ερευνητικό. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην Ευρώπη τι είδους παρέμβαση, επέμβαση κατά των εγκληματικών οργανώσεων. Παίρνοντας περισσότερο το γαλλικό μοντέλο από το ελληνικό του κ. Κόρκοραν. Τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιταχθούμε στη μαφία και να γίνει σημείο αναφοράς και για άλλες χώρες. Ευχαριστώ και τους δύο για την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κ. Χάνκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Κολομ... Ο κύριος Κολόμπι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μας εξήγησε ότι στη Γαλλία ε, είναι έχει πολλαπλές εκφάνσεις. Η οργανωμένη εγκληματικότητα μας μίλησε για την ε, ρωσική μαφία, ρωσόφωνη φωνία. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα, ε, καθότι προέρχομαι από την Ουγγαρία και μετά την ε, εξαφάνιση των κομμουνιστικών καθεστώτων παρατηρείται την ε, κεντρική Ευρώπη ένα φαινόμενο που προσωμιάζει το Ιταλικό. Υπάρχουν επίσης ε, με διακλαδώσεις ε, που ενώνουν κρατικές υπηρεσίες με την μαφία. Πρόκειται για εγκληματικέ δραστηριότητες όπως εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να σας περιγράψω τη δράση της ρωσική μαφίας, αλλά μπορώ να σας πω ότι ε, διείσδησε η μαφία ε, στο κράτος ε, της Ουγγαρίας. Αυτό ισχύει για πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, για την Ελβετία, για τη ΣΥΠΑ, ε, παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα και στις τράπεζες ε, τώρα πια δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων περισσότερο από ότι ε, στο εμπόριο όπλων. Σας ρωτώ λοιπόν, στη Γαλλία μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν, υπάρχει ακόμη ρωσική μαφία. Ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κόρκοραν είναι παρόν κατόπιν δική μου ουσιαστικά παρέμβαση. Χαίρομαι που είναι εδώ, διότι κάποιοι που δεν είχαν ε, πόρου φανερούς ζούσαν σαν εκατομμυριούχοι. Και άλλοι που ήταν στο επίδομα ανεργία είχαν ε, δύο-τρία σπίτια. Και ο κόσμο βαρέθηκε να τα βλέπει αυτά. Και η κοινή γνώμη πραγματικά θέλει να βλέπει να πληρώνει το τίμημα εγκληματίε. Αυτό είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να μάθουμε και το εφαρμόσουμε σε όλη την Ευρώπη αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα που μας παρετέθη. Δύο ερωτήσει. προς τον κύριο Κόρκοραν. Πρώτον, το αστικό δίκαιο χρησιμοποιείται, όχι το ποινικό, έτσι. Δεν χρειάζεται να θεωρηθεί ένοχος για ποινικό αδίκημα κάποιος. Βάσει πιθανότητων σταθμίζει το δικαστήριο. Πώς γίνεται, χρησιμοποιείται αστικό δίκαιο πριν έχει αποδειχτεί διάπραξη εγκλήματος. Δεύτερον, Όσον αφορά την απόφαση δικαστού Μαγκίνης, όσον αφορά την ισορροπία των δικαιωμάτων, δεν θέλανε να δώσουν στους ανθρώπους των εισοδήματος, να συνεργαστούμε στο και κλπ, διότι είχαν ιδιωτικές πληροφορίες, η Πώς μπορείς να καταδιώξεις αυτούς τους εγκληματίες, αλλά να μην παραβιάσεις τα δικαιώματα των ομίμων, ε, των ομοταγών πολιτών ε, με τη χρήση ε, εμπιστευτικών πληροφοριών. Η δικαστή Μαγκίνε αποφάσισε ότι υπήρχε αυτή η ισορροπία, η σωστή ισορροπία. Μήπω μπορείτε να πείτε περισσότερα όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Κοστέλο, για ένα λεπτό, κυρία Κοστέλο. Συγγνώμη Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές και από τις τρεις χώρες για τις παρουσιάσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν. Προ τον ε, κύριο Κόρκοραν. Η παρουσίασή σα ήταν άκρο ενδιαφέρουσα. Γνωρίζω και καλύτερα την κατάσταση στην Ιρλανδία. Κάποιε ερωτήσει: Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται, είπατε ότι 7 χρόνια περνάνε πριν μπουν ξανά στο σύστημα. Προσπαθούσα να κάνω εξατία λέγοντα ότι τα έσοδα, ένα ποσοστό των εσόδων αυτών θα έπρεπε να μπαίνει στην άκρη για να ξαναμπούν στην ε, κοινωνία, σε Κίνους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Και είναι κυρίω ε, ε, οι, προβληματικοί άνθρωποι, ε, όπως τα ναρκωτικά έχουν δημιουργήσει αυτές τις κοινότητες μεγάλα προβλήματα. Έχετε σκεφτεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2012 ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νέα οδηγία. Παρόμοιο αυτό που κάνουμε στην Ιρλανδία χωρίς πρώτερη καταδίκη. Έχουμε δυνατότητα αυτοεξαίρεσης στην Ιρλανδία όσον αφορά τις οδηγίες. Πώς μπορούμε να ενταχθούμε αντίθετα, αντί opt-out, να κάνουμε opt-in στην οδηγία. Και τι εμπόδια υπάρχουν. Ερώτηση για όλους. Συλλογή στοιχείων. Πρόσβαση στα αρχεία στοιχείων κινητών τηλεφώνων και τα στοιχεία διατηρούνται πάνω από ένα εξάμεινο. Όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο, τι είδα. Πολλοί εγκληματίε χρησιμοποιούν μη καταχωρημένα κινητά. Άρα δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία για αυτά τα κινητά. Μπορούμε να υποχρεώσουμε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να καταχωρούν τους αριθμούς κινητών και να υπάρχει και κάποια δυνατότητα ανιχνευσιμότητας. Γετόβα. Γιώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, όλους τους ομιλητές ε, του απογεύματο. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι παρουσιάσεις. Έχω πολύ ιδιαίτερη ερώτηση εγώ στον κύριο Κόρκορα. Αν κατάλαβα καλά, εσείς τροποποίησατε τη νομοθεσία σας το καλοκαίρι του 1996 και για την κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος πλέον δεν χρειάζεστε πρώτερη ποινική καταδίκη. Επειδή τώρα ε, εκπονούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω τι λέει η πρακτική σας εμπειρία. Ε, αυτή η νομοθεσία ε, δίνει έδαφος για καταχρήσεις και για πολιτικοποίηση του όλου θέματος. Ασκούνται πολιτικές πιέσεις σε ορισμένους εκπροσώπους επιχειρηματικού κόσμου. Βάιλερ, για κάτι διαδικαστικό θέλετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, μια τεχνική ερώτηση, διαδικαστική. Και ο συνάδελφος εδώ παρακαθήμενος. Τον τελευταίο μιλητή δεν θα τον ακούσουμε και θα συζητήσουμε. Το 12, δεν ξέρω, είπατε τίποτα στην αρχή της συνεδρίασης και δεν το πήραμε είδηση. Ναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο και ενδιαφέρον τι θα κάνουμε, θα το αναβάλουμε για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ehm, Όπως σας είπα, συσσωρεύσαμε μεγάλη καθυστέρηση. Και στην ερώτηση που κάνατε, τι να κάνω, να ζητήσω τον κύριο Κολομπή και τον κύριο Κορά να στείλουν γραπτό ή δυνατόν τι απαντήσει, διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να μην του ακούσουμε. Να μην ακούσουμε την παρέμβαση του Προέδρου Λατόρε, και δεν το θεωρώ σωστό. Να δώσω αμέσως το λόγο στον πρόεδρο Λατόρα, πρόεδρο του Δικτύου Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι κινητήρα για κάθε σοβαρή απόφαση που λαμβάνεται σε πολιτικό επίπεδο. Σας δίνω αμέσως το λόγο και ε, να έχετε υπόψη το δίκτυο FLAIR που είναι δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών που αντι... αντιτάσσεται στο διεθνές οργανωμένο εγκλήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκληση να συνεργαστούμε και να συμμετάσχουμε στις εργασίες της Επιτροπής σας. Ελπίζω πραγματικά οι προσδοκίες σας ε, να μην ε, αποδειχθούν φρούδες. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά συστήθηκε αυτή η Επιτροπή. Οπότε εγκρίναμε τότε την, ε, τον νόμο Λατόρε που για πρώτη φορά ε, θέσπισε το, στον ποινικό κώδικα ε, και έκανε αδίκημα την σύσταση συμμορία με σκοπούς τύπου μαφίας και επίσης να κατάσχονται τα προϊόντα του εγκλήματο και μέτρα προληπτικά που είχαν σαν στόχο να πλήξουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Ο πιο τώρα, ο πατέρας μου που ήταν βουλευτή και συνέταξε το νόμο που έχει το όνομά του δεν μπόρεσε να δει την έγκριση του το Σεπτέμβριο του 1982 διότι σκοτώθηκε από τη μαφία στις 30 Απριλίου του χρόνου αυτού, αυτού. Ένας νόμος που όπως είπε και ο εισαγγελέο ο κ. Γκράσο που η διεθνή κοινότης ε, θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το ΦΛΕΡ, το δίκτυο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και το οποίο να προεδρεύω, ε, διαδέχεται, το, διαδέχεται το δίκτυο του Λίμπερα που ήθελε να εφαρμόσει τις αρχές της ελευθερίας και τη πολιτισμική αντίσταση και τη κοινωνική αντίσταση ε, κατά των εγκληματικών αυτών οργανώσεων. Το Λίμπερα το 1996 πρωταγωνίστησε σε μια έκτακτη εξαιρετική κινητοποίηση λαϊκή και συνελέγησαν ένα εκατομμύριο υπογραφέ για υποστήριξη για την κοινωνική χρήση των κατασκευέντων περιουσιακών στοιχείων. Μια πρωτοβουλία από το Κοινοβουλίο εκείνο τον ίδιο χρόνο ε, θέσπισε μέσω νομοθεσία. Εισήγαγε σε νόμο. Το Φλερ ιδρύθηκε το 2009 και σε αυτό εδώ το κτίριο Ιδρύθηκε λέγω το 2009 το ΦΛΕΡ, αξιότιμοι βουλευτές, σε μια συνέλευση που έλαβε χώρα εδώ, στη Μικύκλιο, σε αυτό το κτίριο, όπου εσείς εκεί ασκείτε ε, το νομοθετικό σας έργο και την εξουσία σας. 47 ενός Ευρωπαϊκής Ενώσης εκπροσωπεί της πρώην Ιουγκοσλαβίας, της Ανατολικής Ευρώπης, της περιφερικής του Κάφκασου και της Μεσογειακής Λεκάνης. Οργανώσει που θέλουν να αντιτάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα. Συγγνώμη πρόεδρε, διακόπτη Πρόεδρε. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Θέλει να μιλήσει ο κύριος Τόρε. Άρα ε, περίμενε πάνω από τη τέταρτα της ώρας όποιος ενδιαφέρεται ας φύγει από την αίθουσα να επιτρέψουμε στον πρόεδρο να κάνει την ομιλία του, την παρουσίασή του. Επιτρέπετε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο Έλεγα λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, ότι το φλερ στις διάφορες χώρες και σε διεθνές επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί προγράμματα δραστηριοποίησης, ε, προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης που απευθύνεται κυρίως προς τις νέες γενιές δεν, δεν θέλουμε να παραθέσουμε όλες τις πρωτοβουλίες που ακολουθήσαμε τις, τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας μας. Αν θέλετε μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας www.flair.net Να υπενθυμίσω μία από τις πρωτοβουλίες και είμαστε ιδιαίτερη υπερήφανοι για αυτή. Όλε, ε, σημαίνει ε, πέρα από την νομιμότητα στην Ευρώπη. Το Summer School, το Summer Camp, το Youth Forum ε, για τρίτη χρονιά θα οργανώσουμε τέλος Ιουλίου στην περιοχή της Πούλια, στην Νότια Ιταλία, με τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων από όλη την Ευρώπη και με πολλούς επιφανείς ειδικού σε εθνές επίπεδο για να μελετήσουμε και να εμβαθύνουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες όσον αφορά το θέμα της νομιμότητας και του οργανωμένου εγκλήματος σε διεθνές επίπεδο και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των νέων στην Ευρώπη που γνωρίζει το πόσο επικίνδυνο είναι το οργανωμένο έγκλημα και οι σχετικέ οργανώσει πόσο μπορούν να δυσδύουν και στην καθημερινή μα ζωή. Ε, νέοι που δεσμεύονται καθημερινά να κάνουν μάχε σε πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο ούτω ώστε η μαφία να μην επηρεάσει το μέλλον του. Το φλερ επενδύει πάνω του κυρίω, διότι θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σε μία μάχη που εμεί οι ενήλικε ακόμα δεν καταφέραμε να νικήσουμε, να κερδίσουμε. Φέτο είναι η χρονιά όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση οδηγία όσον αφορά την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματο σε υποέγκριση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπαίνω τώρα στην ουσία αυτού του νομοθετήματο. Κλείνω λέγοντα ότι για μα αντιπροσωπεύει μια νέα πρόκληση. Διότι όπω το φλερ θέλουμε να διαδώσουμε και να γνωστοποιήσουμε στου πολίτε, άντρε και γυναίκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλε τι χώρε, αυτό το εργαλείο του ΦΛΕΡ που είναι ένα μέσο καταπολέμησης ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ εσάς κύριε Πρόεδρε, κύριε Λατόρε για την συνεισφορά σας κυρίως όσον αφορά ε, την χρήση αυτών ε, των προϊόντων για κοινωνικούς σκοπούς. Δίνω το λόγο στους συντονιστές. Κυρία Μάτια έχει το λόγο για το καταρχάς. Σα ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας σε αυτόν τον δύσκολο ομολογουμένο αγώνα. Θα ήθελα να μας πείτε ή δυνατόν αν υπάρχουν νέοι σε κάποιες χώρες που εμπλέκονται περισσότερο στην καταπολέμηση. Ε, στο Βορρά, παραδείγματο χάρη, υπάρχει συνήθω μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων σε σχέση με τον Νότο ή το αντίστροφο. Εσείς τι εμπειρία έχετε, υπάρχει κάποιο κοινωνικό μοντέλο συμμετοχής, σε ποια κράτη συμμετέχουν περισσότερο είναι... Ε, Κύριε Φαγιόν, η κύριε Μπορσελίνο. Ναι, έχω μόνο μία παρατήρηση να κάνω. Χαιρετίζω με ευχαρίστηση τον Φράνκο Λατόρε και θα ήθελα να υπενθυμίσω ως αντιπρόεδρος της Λίμπερα το 1996 Ήρθαμε το Λουίτζι Σότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρουσιάζαμε την ένωση αυτή, τη Λίμπερα, την οργάνωση αυτή. Και θυμάμαι ότι έλεγαν ότι δεν υπήρχε πουθενά αλλού στην Ευρώπη ένα συντονισμό οργανώσεων που είχα σαν στόχο την καταπολέμηση της μαφίας και την προώθηση της ε, κοινωνίας. Και υπήρξε πολύ ενδιαφέρον πλευράς διαφόρων βουλευτών και η Ένωση Φλερ είναι η υλοποίηση εκείνου που τότε φαινόταν μόνο ένα όνειρο και, κάτι, και παράξενο όνειρο και να το βλέπω αυτό με κάνει να σκέφτομαι και να υπογραμμίζω ότι πράγματι όταν κανείς προσπαθεί να προωθήσει κάτι και κάτι το οποίο φαίνεται αδύνατο τελικά φτάνουν τα αποτελέσματα και νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει καθημερινά το Φλερ. Σας ευχαριστώ λέει πρόεδρος εκτός μικροφών. Ο κύριος Νιούτον Ντόν έχει το λόγο για ένα λεπτό συντομία, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αναρωτιέμαι, ε, ε, έρχονται πολλοί νέοι από το δικό μου κράτος, ε, στο βορρά της Ένωσης. Και αναρωτιέμαι γιατί είσαστε στη Νότια Ιταλία, γιατί εκεί οργανώνει τι εκδηλώσει, ενώ είναι η καρδιά του οργανωμένου εγκλήματο. Μήπω του βάλετε στον πειρασμό να στρατολογήσουν του νέου σα και του μαφιόζου. Κύριε Λυπάμαι τώρα που έχουμε τόσο λίγο χρόνο για αυτό τόσο σημαντικό θέμα. Ή τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Ε, ποιες δυνατότητες έχουμε να ενισχύσουμε δεχομένω την ευρωπαϊκή διάσταση ε, αυτού του θέματος, δηλαδή να κάνουμε περισσότερους νέους να ενδιαφερθούν. Ευχαριστώ. Λυπάμαι και εγώ που έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θα πρότεινα η συνεδρίαση των συντονιστών που αργο... στη συνεδρίαση των συντονιστών που προβλέπεται αργότερα να ξανακούσουμε τον το Φλερ και τον πρόεδρο κύριο Λατόρε ε, ε, όταν έχουν περισσότερη ηρεμία. Ε, διότι περιοριστήκαμε σε πολύ ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά σωρεύσαμε καθυστέρηση μεγάλη. Και εγώ λέω ότι δεν μου αρέσει να λέω κομπλιμέντα διότι δεν πρόκειται όμως για κομπλιμέντα εδώ. Ε, εσείς σημειώσατε και σημειώνετε όχι μόνο στην Ιταλία. Ε, είστε ένα παράδειγμα κι αλλού. Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαν ε, για σας. Ε, σ' άλλο βήμα που συζητούσαμε και σας θέσαμε εσά σαν παράδειγμα προς μίμηση. Διότι κάποιοι εκπρόσωποι διαφόρων χωρών στη συνάντηση αυτή είπαν ότι τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ε, είναι καλύτερο να απολούνται, να δίνονται ε, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα για τις χώρες που κάνουν την κατάσχεση. Αλλά το δικό σας παράδειγμα είναι προς μίμηση. Σας ευχαριστώ για το πάθος με το οποίο καθημερινά εργάζεστε, αλλά δεν είναι μόνο πάθος. Είναι κάτι που υπάρχει αυτό στο ίδιο το γενετικό σας υλικό, στο DNA σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη Είπατε, εγώ μπορώ να, όπως κάνετε στο προηγούμενο, μπορώ να απαντήσω γραπτό στις ερωτήσεις που μετέθησαν από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ εσάς, Πρόεδρε Λατόρε. Και τώρα ξεκινάμε αμέσως τη συνεδρίαση των συντονιστών που υπενθυμίζω γίνεται κυκλισμένων των θυρών.